Καλησπέρα σας. Άρχεται η συνεδρίαση της Επιτροπής Μεταφορών. Έχετε ενώπιον σας ε, το σχέδιο μερίσιας διάταξης για το διήμερο που μας περιμένει. Δεν ξέρω αν είστε ικανοποιημένοι όλοι. Ωραία, σας ευχαριστώ. Στη συνέχεια έχουμε την έγκριση των πρακτικών ερωτήσεις για τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης. Αν όχι, μπορούμε να εγκρίνουμε τα πρακτικά. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Κατόπιν έχουμε το πρώτο σιδηροδρομικό πακέτο. Ε, θα συζητήσουμε τις τροπολογίες. Η εισηγήτρια είναι η κυρία Σερακιάνη. Κυρία Σερακιάνη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να παρουσιάσω λίγο στην Επιτροπή μας ε, το πώς έχει η κατάσταση των εργασιών μας. Με τους κοιόδης εισηγητές ε, συζητήσαμε κάποιες συμβιβαστικές ε, δυνατότητες για κάποια βασικά θέματα της αναδιατύπωσης, κυρίως για το ρυθμιστικό φορέα, για τη χρηματοδότηση, για τις πράξεις κατεξουσιοδότηση και για το άρθρο 13. Όσον αφορά το ρυθμιστή υπάρχει συμφωνία ε, ο ρυθμιστής θα είναι υπεύθυνο για την εποπτεία και θα ε, πρέπει να ε, εποπτεύει ώστε να μην υπάρχουν διακρίσεις και να αποφεύγονται. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ρύθμισης θα ορίζονται βάσει των αρμοδίων εθνικών κοινοβολέων ή των αρμοδίων κοινοβουλίων και θα πρέπει να υπάρχει και δήλωση οικονομικών συμφερόντων, να είναι ανεξάρτητη και δεν θα πρέπει να επηρεάζονται σε καμία περίπτωση από την κυβέρνηση ή από κάποια ιδιωτική ή δημόσια επιχείρηση. Οι ρυθμιστές ε, λαμβάνουν ε, αποφάσεις και δρούν με ίδια πρωτοβουλία για να ρυθμίσουν σε ένα μήνα αφότου δεχτούν ένα αίτημα ε, διαθέτης κάποιου ζητήματος. Επίσης, αν υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει καταγγείλει διακριτική συμπεριφορά, μέσα σε δύο εβδομάδες ε, η Επιτροπή, αν είναι απαραίτητο, θα ζητά να γίνουν όλες οι αλλαγές. Από τότε ε, η περίοδος του ενός μηνός θα παρατείνεται για ένα μήνα επιπλέον. Θα πρέπει επίσης να γίνεται ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνιστών για τις δραστηριότητές τους και θελήσαμε να ε, επισημάνουμε την ενίσχυση του εθνικού ρυθμιστή, αλλά επίσης να δημιουργήσουμε απευθείας και ένα δίκτυο μεταξύ των εθνικών ρυθμιστών ώστε να δίνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τις δραστηριότητές τους, ένα δίκτυο το οποίο επισήμως θα πρέπει να συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα κατόπιν προσκλήσεως της Επιτροπής. Και ε, γι' αυτόν ακριβώς το σκοπό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει ότι θα υπάρχει και ενεργός συνεργασία μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών και να παρεμβαίνει εάν οι ρυθμιστικές αρχές δεν μπορούν να πληριώσουν τις ε, υποχρεώσεις τους. Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να δημιουργήσει δημιουργήσει και μία τράπεζα δεδομένων, μία βάση δεδομένων όπου θα δίνονται όλα τα στοιχεία των αιτήσεων, ε, να δίνονται ημερομηνίε, η έναρξη διαδικασίας, οι τελικές αποφάσεις, ε, τα συμβαλόμενα μέρη, ε, τα βασικά ζητήματα που αφορούν πρόσβαση και κόστος ε, διεθνικών ε, σιδηροδρομικών υπηρεσιών. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τον ε, εθνικό ρυθμιστή. Όσον αφορά τώρα το θέμα της χρηματοδότησης, προβλέποντας εδώ κάποια πράγματα, θα πρέπει να υπάρχουν κάποια προγράμματα επενδύσεων και να διασφαλίσουν ότι θα ε, γίνεται διαβούλευση πριν εγκριθεί το επιχειρηματικό σχέδιο. Τα κράτη-μέλη από πλευρά του θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι ο διαχειριστή του συστήματο δεν θα έχει έλλειμμα χρηματοδότηση για δύο συνεχή χρόνια και θα πρέπει να υπάρχει και μια ισορροπία αφενός ε, τα όσα προέρχονται από άλλες εμπορικές δραστηριότητες και κρατικά κονδύλια και αφετέρου το κόστος των υποδομών συμπεριλαμβανομένων και των προβλεπόμενων ε, ε, δαπανών για τις ε, πολιετής δαπάνες και την αηφόρα ανάπτυξη. Για το άρθρο 13 τώρα, ένα άρθρο που συζητήσαμε στην τελευταία συνεδρίαση που είχαμε με τους κοιόδης εισηγητές, Έχουμε μια συμβιβαστική πρόταση στην οποία προβλέπεται η χωρίς διάκριση πρόσβαση από όλους τους διαχειριστές υποδομών καθώς επίσης και ε, το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση σε όλες τις σιδηροδρομικές υπηρεσίες και στις ε, ε γραμμές ε, βάση του κανονισμού. Ε, θα πρέπει να υπάρχει και ένα σταθερό χρονικό διάστημα το οποίο θα καθορίζεται από τον εθνικό ρυθμιστή που θα δίνει τη δυνατότητα σε τεχνικές υπηρεσίες. Εάν υπάρχει άρνηση πρόσβασης στις υπηρεσίες ο διαχειριστής θα πρέπει να προσφέρει μια εναλλακτική λύση η οποία θα είναι τεχνικός και οικονομικός ε, εφικτή χωρίς ε, να υπάρχει ουσιαστική αύξηση του κόστους. Εάν δεν μπορούμε να βρούμε εναλλακτική λύση, τότε ο ρυθμιστής θα πρέπει να αναλάβει όλα τα μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες των ενδιαφερομένων. Τέλος, εάν ε, ένα κέντρο βοήθειας δεν έχει χρησιμοποιηθεί για τουλάχιστον ένα έτος, θα μπορεί να χρησιμοποιεί για εναλλακτικές δραστηριότητες του σιδηροδρομικού τομέα, εκτός και αν αποδεικθεί ότι υπάρχει μια διαδικασία μετατροπής που δεν επιτρέπει τη χρήση από τη σιδηροδρομική υπηρεσία. Αυτά είναι λοιπόν τα τρία ζητήματα ε, για τα οποία έγινε μια συζήτηση. Σε αυτά προσθέτουμε και τις πράξεις κατεξουσιοδότηση και έγιναν κάποιες προτάσεις συμβιβαστικές και υπήρξε και η συζήτηση με τους κοιόδης εισηγητές μετά από τη συνεδρίαση της Επιτροπής μας θα γίνει και συνεδρίαση και πάλι με τους κοιόδης εισηγητές και θα συζητήσουμε τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με το παράρτημα 3, με το άρθρο 30 και το παράρτημα 7, τα άρθρα 31 και 32 και το παράρτημα 8, το άρθρο 15 παράρτημα 1, τα 6 και 7 με το παράρτημα 1α και επίσης θα γίνει και συζήτηση για τις τροπολογίες που σχετίζονται με το άνοιγμα της αγοράς. Αυτά όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα των εργασιών μας. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, Mr. Kuhn, for the PPE. Danke, Herr Vorsitzender. Danke auch an die Berichterstatterin, Frau Seracani. Es hat sich natürlich herausgestellt, dass das ein sehr wichtiges Thema ist Ευχαριστώ πολύ. Από ό,τι φαίνεται είναι πάρα πολύ ε, ευρύ το θέμα του άνοιγματος των ευρωπαϊκών συνδρομικών αγορών και υπάρχουν και πάρα πολλές πτυχές που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ούτως ώστε να βρεθούν πρακτικές λύσεις. Δεν ε, θα επαναλάβω όλα όσα ήδη πολύ σωστά μας είπε η συγγήτρια. Επί του παρόντος βρισκόμαστε στη μέση της όλης διαδικασίας και Υπάρχει αρκετά η προσέγγιση, σύγκληση απόψεων σε ό,τι αφορά τη κατεξουσιοδότηση πράξη, τι δυνατότητε χρηματοδότηση, τα κράτη-μέλη, τι εθνικέ αρχέ. Όλα αυτά τα θέματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Είναι μάλιστα θέματα τα οποία θα είναι και σημαντικά για τη δημιουργία πρόσβασης ε, στην αγορά για όλους ε, τους ε, φορείς εκμετάλλευσης. Είναι πολύ σημαντικό οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές να μην φορταθούν υπερβολικά με διάφορες αποστολές και διάφορα καθήκοντα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει εστίαση ξεκάθαρη πρώτα απ' όλα στην επαλήθευση των τιμών και των συστημάτων τιμών στο επίπεδο των τιμών, διάρθρωση κόστους, πάγια και μεταβλητά έξοδα υποδομές, κόστος και βέβαια σύστημα τιμών για τη χρήση των εργαστηρίων. Κάτι πολύ σημαντικό. Πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και να είναι η ίδια τα κριτήρια για όλους τους φορείς εκμετάλλευσης. Επίσης, διάθεση καυσίμων και εκεί θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη όρη για όλους. Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα έχει να κάνει με την πρόσβαση. Ποια σιδηροδρομική επιχείρηση έχει πρόσβαση στις ευρωπαϊκές αγορές. Μιλάμε για την αδειοδότηση των σιδηροδρομικών εταιριών. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και θα πρέπει να εφαρμόζονται κριτήρια για τη συμμετοχή στην αγορά. Ήδη όμως ε, παρατηρούμε μεγάλη καθυστέρηση. Δύο χρόνια δεν έχουμε καταφέρει τίποτα. Θα πρέπει εντός έξι μηνών να έχουμε προχωρήσει, πρέπει να το συζητήσουμε και πρέπει να συνεργαστούμε και με τις εθνικές ε, ε, αρχές ασφαλείας οι οποίες θα πρέπει επίσης να, συμβάσουν, να συμβάλλουν σχετικά με, τις, ε, ε, με τους οργανισμούς υπηρεσιών. Ε, εκεί υπάρχει συνήθως το πρόβλημα και δεν θα τα καταφέρουμε ε, διότι εάν εδώ απλούστατα λέμε ότι ε, ένας ε, ένα σιδηρόδρομος δεν χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις και πρέπει αυτές να διατεθούν στην αγορά θα είναι μια δύσκολη διαδικασία διότι θα δυσχεράνει την κατάσταση των ενδιαφερομένων διότι αυτό που είναι σημαντικό είναι πόσο καιρό πρέπει να, ε, επενδύουν οι σιδηρόδρομοι για να μπορέσουν να ε, υπάρξει μία συγκεκριμένη εγκατάσταση διότι όσον αφορά το Και γι' αυτό σχετικά με την με την πολιτική μου ομάδα το ΕΛΚ θα είναι δύσκολο να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση διότι υπάρχουν διάφοροι κανόνες οι οποίοι εμπλέκονται και ιδίω η μεταφορά μεταξύ ε, του οργανισμού και του διοικητού των σιδηροδρόμων θα πρέπει να υπάρχει ε, διαφάνεια, να ξέρουμε ε, τι αμείβεται ο κάθε ένας και θα πρέπει να γνωρίζουμε ε, τι είναι οι παροχές που προσφέρουν τα κράτη-μέλη στις οργανώσεις τους και να δούμε πώς θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα κοινό πόρισμα χωρίς να επισέλθουμε σε λεπτομέρειες και όσον αφορά το unbundling το οποίο μπορεί να θεωρηθεί σαν μία λύση θα πρέπει να μην θεωρηθεί ότι είναι κάτι τελείως ανόητο και αν μπορέσει να προχωρήσει. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον ο Στέρκερχη Στέρκ τώρα τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εκπροσωπώ τον ε, συνάδελφο Ραμός, ο οποίος είναι σκιώδης εισηγητής δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειες, γιατί μεταξύ των εισηγητών και μάλλον των σκιωδών εισηγητών στις συνεδρίες θα τα πει ο ίδιος μόνος του. Απλά να σας παρουσιάσω κάποια θέματα αρχής, σημαντικά για μένα και για την ομάδα. Πρώτα απ' όλα, το θέμα είναι πάνω απ' όλα το άνοιγμα της αγοράς. Αυτό είναι το σημαντικό. Και αυτός είναι ο στόχος που πρέπει να επιδιώξουμε. Το άνοιγμα των αγορών. Επί του παρόντο, η κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ιδεώδη. Θα πρέπει λοιπόν τι προτάσει που έχουμε επιτάπητο να τι αξιοποιήσουμε για να επιτύχουμε το στόχο που ανέφερα, δηλαδή το άνοιγμα των αγορών. Και ξεκινώντα από αυτό, ένα σημαντικό στοιχείο για την ομάδα μου είναι να φροντίσουμε κάθε κράτο μέλο να έχει μια ισχυρή ρυθμιστική αρχή, η οποία θα είναι σε θέση να κρίνει τις σχέσεις μεταξύ των εταιριών που διαχειρίζονται και μεταξύ των ε, συνδρομικών εταιριών, αν υπάρχει διαφάνεια κτλ. Πρέπει να υπάρχει μια αρχή η θα τα εξετάζει αυτά σε κάθε κράτος μέλος. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις συμβαστικές προτάσεις που έχουν υποβληθεί, παρατηρώ ότι είναι κάποια στοιχεία που περιπλέκουν ιδιαίτερα το όλο θέμα και οι περιπλοκές και οι επιπλοκές αυτές θα μειώσουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα των εθνικών ρυθμιστικών αρχών. Παραδείγματο χάρη συμβαστική πρόταση 56-3C που λέει ότι θα ε, αναφέρει η Εθνική Ρυθμιστική Αρχή στην Κομισιόν όλε τι προτάσει κτλ. Και, και μετά αναφέρονται όλε οι παράγραφοι. Και σε δύο εβδομάδε ε, θα ζητήσει ε, ενδεχομένως η Κομισιόν να γίνουν κάποιες τερθωτικές κινήσεις. Μα πρέπει να πούμε ότι έχουμε 27 ρυθμιστικές αρχές, οι οποίες θα πρέπει να υποβάλουν όλες τις προτάσεις απόφασής τους στην Κομισιόν που θα πρέπει να συμφωνήσει να μην συμφωνήσει μέσα σε δύο εβδομάδες. Καταλαβαίνετε τι πρόκειται να γίνει. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Και δεν έχει κανένα, ε, καμία δυνατότητα να πετύχει αυτό το, το πράγμα. Είναι λίγο απλουστευτικό το όλο. Ε, θέμα. Δεν νομίζω ότι ουσιαστικά όμως οδηγεί ε, σε πραγματική απλούστευση, ούτε ενισχύει τις αρμοδιότητες των εθνικών ρυθμιστικών αρχών. Αν υπάρχουν, μια, αν υπάρχουν εθνικές ρυθμιστικές αρχές που έχουν ε, κάποια δύναμη, δεν ξέρω μήπως θα ήταν καλύτερο αντί της Κομισιόν να έχουμε μια ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή. Αλλά δεν υπάρχει. Αυτό τέλος πάντων σταδιακά προχωράμε το θέμα είναι η Κομισιόν να μην είναι μια δεύτερη διοίκηση που θα πρέπει να τα παληθεύει όλα, απλά να είναι ένα είδος ε, οργανισμού προσφυγής. Το θέμα είναι να, υπάρχει αποτελεσματικότητα. Ε, σε ό,τι με αφορά, όπως είπε και ο συνάδελφος Κούν, είναι προφανές ότι η Εθνική Ρυθμιστική Αρχή θα πρέπει να φροντίζει να υπάρξει διαφάνεια. Σε ό,τι αφορά τώρα τη σχέση μεταξύ διαχειριστών και ε, συνδρομικών εταιριών, η Εθνική Ρυθμιστική Αρχή θα πρέπει να φροντίσει οποιαδήποτε κίνηση ποσών, χρηματικών ποσών να γίνεται με διαφάνεια και να είναι ξεκάθαρη και δεν θα, υπάρξει, δεν θα πρέπει να υπάρχουν προνομιακέ σχέσει μεταξύ διαχειριστών υποδομών και συνδρομικών εταιριών. Αυτό θα πρέπει να επιβλέπουν οι εθνικέ Ρυθμιστικέ αρχέ. Μία τελευταία παρατήρηση κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει ε, ακόμη ε, κάποια προσπάθεια απλούστευσης. Η ομάδα μας έχει ε, την άποψη ότι επιδέχεται η πρόταση ακόμη κάποιες απλουστεύσεις. Και να σας πω ότι θα πρέπει όλοι να σκεφτούμε τις επιπτώσεις του άρθρου 8 επί της χρηματοδότησης του διαχειριστή υποδομών. Τα κράτη-μέλη ουσιαστικά πρέπει να διαβουλεύονται με όλους, με όλο τον κόσμο πριν υποβάλει το στρατηγικό σχέδιο που πρέπει να υποβάλει για τις υποδομές του. Πριν το κάνει αυτό πρέπει να ε, έχει συνεννοήσεις με όλους, τοπικές αρχές, περιφερειακές αρχές, διάφοροι stakeholders, όπως λέμε, εμπλεκόμενοι φορείς, συνδικάτα και όχι μόνο ε, τα γενικά αλλά και τα τομεακά, τα, τα, κλαδικά ε, και εγώ δεν ξέρω ποιον άλλο. Πότε θα ολοκληρωθεί λοιπόν αυτό το στρατηγικό σχέδιο. Ήδη στη δική μου χώρα δεν είναι εύκολο ε, το να λαμβάνονται αποφάσεις, αλλά χρειάζονται διαβουλεύσεις με όλους. Όταν θα έχουμε φτιάξει αυτό το στρατηγικό μας σχέδιο, δεν θα υπάρχουν πια σιδηρόδρομοι, στη χώρα μου τουλάχιστον. Το θέμα είναι, επαναλαμβάνω, υπάρχει αποτελεσματικότητα πάνω απ' όλα. Αυτός είναι ο στόχος. Και λέει για τα κράτη-μέλη που πρέπει να παρέχουν χρηματοδότηση ε, στον ε, διαχειριστή υποδομών. Στα αγγλικά χρησιμοποιείται η λέξη shall. Παρέχουν χρηματοδότηση. Δηλαδή, ό,τι και να κάνει ο διαχειριστής υποδομών, το κράτος θα πληρώσει. Και αν δεν υπάρχουν χρήματα, θα πληρώσει το κράτος. Όλοι ξέρουμε ότι αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει. Ας μην το γράψουμε και στην οδηγία. Όλα αυτά τα λέω για να σας πω ότι όταν διαβάζω τη συμβαστική πρόταση βλέπω και πιστεύω ότι υπάρχουν ακόμη πράγματα τα οποία χρήζουν απλούστευσης. Επίσης υπάρχουν κάποιες διατάξεις επί των οποίων θα πρέπει πραγματικά να σκεφτούμε και να σκεφτούμε τι επιπτώσεις θα μπορούσαν να έχουν. Τέλος, θα ήθελα κύριε Πρόεδρε να επιστήσω την προσοχή σας. Έχουμε την απαιτούμενη συνοχή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συγκεκριμένα στην Επιτροπή μας, ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το θέμα από τεχνικής πλευράς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο όλα να διαρθρωθούν μεταξύ τους και από το α έως το ω να είναι όλα ε, ξεκάθαρα, απλά και όλοι να τα αντιλαμβάνονται. Η σχέση ε, μεταξύ άρθρων, ε, παραρτημάτων, διαφάνεια είναι πάρα πολύ πολύπλοκο θέμα. Νομίζω λοιπόν ότι δεδομένου του τρόπου με τον οποίο εξελίσσεται η συζήτηση αυτή τη στιγμή, δεν είναι δεδομένο ότι υπάρχει αυτή η συνοχή, αυτή η συνεκτικότητα. Αντιθέτως θα έλεγα. Υπάρχει κάποια δυσπιστία μεταξύ, όχι τόσο μεταξύ πολιτικών ομάδων, αλλά και μεταξύ μελών της ίδιας πολιτικής ομάδας. Άρα, ποια είναι η πρώτη μας αποστολή. Απλούστευση και δεύτερη αποστολή, συνοχή, συνεκτικότητα. Εάν η Επιτροπή μας δεν καταφέρει να εκπονήσει ένα συνεκτικό, συνεπές κείμενο, ένα φάκελο που δεν θα έχει εσωτερικέ αντιφάσεις, που είναι δύσκολο γιατί υπάρχουν πολλές παγίδες θα έλεγα σε αυτό το θέμα, τότε θα ε, οδηγηθούμε στην καταστροφή. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας. Βαντάμ. Eh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και για μένα Είναι σημαντικό το θέμα. Θα μιλήσω εκ μέρους ε, του σκιώδους εισηγητού και ε, κατόπιν θα σας πω κάποια δικά μου ζητήματα. Συζητάμε τη δημιουργία ουσιαστικά μιας νέας υπηρεσίας ε, στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν όχι, εμείς διαφωνούμε, ε, διότι εμείς δεν θέλουμε νέα υπηρεσία πηγαίνουμε πολύ μακριά. Όσον αφορά τώρα τη συνεργασία με τις σιδηροδρομικές υπηρεσίες ε, ενισχύ, αυτό είναι αυτό το οποίο θα προτιμούσαμε. Σε καμία περίπτωση δεν θα θέλαμε να δημιουργηθεί μια νέα υπηρεσία. Πηγαίνουμε πολύ μακριά. Δεύτερον, θα ήθελα να ζητήσω από την εισηγήτρια από τούδε και στο εξή να προσέξει την ιδιαίτερη κατάσταση των βαλτικών χωρών. Οι βαλτικέ ε, χώρες αντιμετωπίζουν μια μοναδική και πολύ πολύπλοκη κατάσταση. Αναφέρομαι στην Εσθονία, στη Λιθουανία και στη Λετωνία. Είναι λίγοι οι σύνδεσμοι με, προς το νότο, προς τη Βαρσοβία από τις χώρες αυτές. Ουσιαστικά οι, οι, οι κινήσεις είναι προς την Ανατολή. Και εδώ νομίζω ότι ξέρετε όλο ότι μιλάμε για σιδηροδρομικές υπηρεσίες προς τη Ρωσία, την Λευκορωσία, την Ουκρανία και καταλαβαίνετε ότι οι χώρες ε, αυτές έχουν ε, σιδηροδρομικές υπηρεσίες οι οποίες είναι αποκλειστικώς κρατικές. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο λοιπόν να καταπολεμήσουν ε, οι χώρες της Βαλτικής τις σιδηροδρομικές υπηρεσίες της Ρωσίας, της Ουκρανίας και της Λευκορωσίας οι οποίες θα είναι υποκρατικό έλεγχο. Είναι πολύ περίπλοκη κατάσταση για τι βαλτικέ χώρε. Δεν έχω κάποια λύση να σα προτείνω, αλλά νομίζω ότι στη διάρκεια των εργασιών μα για αυτή την οδηγία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την ε, κατάσταση των βαλτικών σιδηροδρομικών εταιριών και δεν αφορά μόνο τι εταιρείε, αλλά και τους διαχειριστέ των ε, υποδομών της Βαλτική. Διότι αν υποχρεωθούν να αυξήσουν τις τιμές τους οι διαχειριστέ ε, των σιδηροδρόμων στη Βαλτική, ε, όσοι ε, κατευθύνονται προς τη Ρωσία θα έχουν κάθε συμφέρον να περάσουν από την Αγία Πετρούπολη και όχι να κατευθυνθούν προς τη Βαλτική. Ε, και αυτό όχι μόνο για τους σιδηροδρόμους αλλά και για σκάφη. Ε, θα ήθελα λοιπόν να σας επιστήσω την προσοχή στο θέμα αυτό και στην εισηγήτρια αλλά και στην Επιτροπή εν γέννη. θα ήθελα να ξέρω και την αντίδραση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί του θέματο. Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ με τον κύριο Στέρξ, ο οποίο λέει ότι ο στόχο του θέματο αυτού είναι η απελευθέρωση, η πρόσβαση τη αγορά και γι' αυτό θα πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε αποτελέσματα. Στη χώρα μου, κάθε φορά που υπάρχουν περισσότερες θέσεις για νέους διαχειριστές υποδομών είναι προς όφελος ε, των καταναλωτών, των επιβατών, των χρηστών. Επομένως θα πρέπει να ακολουθήσουμε τη συγκεκριμένη άγουσα. Βεβαίως δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα. Ε, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τη σχέση μεταξύ μεταφορέων και διαχειριστών ε, των υποδομών. Α, θα πρέπει να γίνει πλήρης αποσύνδεση μεταξύ των δύο. Αποκλείεται οι δύο αυτοί να είναι στην ίδια επιχείρηση. Κατ' εμάς θα πρέπει να γίνει καταμερισμός και θα πρέπει να γίνει και διαχωρισμός όταν συζητάμε για την αύξηση των τιμών. Ο διαχειριστή των υποδομών δεν είναι αρμόδιο για αυτά τα θέματα κατά την άποψή μου. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει πλήρη διαχωρισμό μεταξύ διαχειριστή υποδομών και μεταφορέα. Δεν θα πρέπει ο ένα να μπορεί να ελέγξει την αύξηση των τιμών των, ε, του άλλου. Δεν γίνεται αυτό σε καμία άλλη ε, μορφή μεταφορά. Δεν θα θέλαμε λοιπόν να υπάρχει και στου υδροδρόμου. Γι' αυτό λοιπόν σα ευχαριστώ την προσοχή. Όσον αφορά τώρα τη λειτουργία τη αγορά. Εμείς επιθυμούμε στη συγκεκριμένη πρόταση να υπάρχει και κίνητρο για το μεταφορέα να χρησιμοποιεί πιο καθαρά, ε, πιο οικολογικά τρένα. Θέλουμε λοιπόν να υπάρχει μία διαφοροποίηση ε, όπως για παράδειγμα χρησιμοποιούνται πιο αθόρυβα και πιο καθαρά τραμ, να μπορούν ε, να υπάρχουν και κατάλληλα κίνητρα να χρησιμοποιούνται καλύτερες σιδηρόδρομοι με καλύτερες τιμές. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές τα καθοριστικά στοιχεία για τη συζήτηση και θα ήθελα να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα των βαλτικών χωρών. Ευχαριστούμε κύριος Κούν είπε ότι η απελευθέρωση είναι ένα εκτενές θέμα και εμείς το καταστήσαμε τόσο εκτενές διότι αυτά τα οποία ετοίμασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν αναδιατύπωση από το 2001 ο νόμος ήταν σαφής και επί εννέα χρόνια κοιμότανε και μετά μας ξετρύπωσε. Το θέμα είναι αυτό το οποίο υπάρχει στην Ευρώπη ε, συνάδει με την νομοθεσία του τότε διότι έχει προχωρήσει η πρόοδος και η μη απελευθέρωση των σιδηροδρόμων ο κανόνας. Υπάρχουν λίγες εξαιρέσεις που μπορεί να αποφασίσουμε και ε, τι θα γίνει περαιτέρω θα αποφασιστεί από το δικαστήριο. Αλλά εμείς ε, για τρίτη φορά συζητάμε το θέμα ε, σε γενική σε γενικές γραμμές και αν καταρτίζαμε τις βασικές μας αρχές ε, θα προχωρούσαμε διότι χρειαζόμαστε ε, και συμφωνούμε όλοι ότι θέλουμε να υπάρχει ένας ανεξάρτητος ρυθμιστής ότι θα πρέπει να υπάρξει απελευθέρωση για να υπάρξει ε, πρόοδος και να περιληφθούν και οι ποτάμιες οδοί. Αν είχαμε συμφωνήσει σε όλα αυτά θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε τώρα. Έπρεπε να καθορίσουμε τις προθεσμίες από την αρχή, από την υποδοχή. Δηλαδή να μην μπορεί ο καθένας να ερμηνεύσει το θέμα διαφορετικά. Εάν δηλαδή εγώ θέλω να... Εάν έχω ένα αίτημα πρέπει να μπορώ να απαντήσω εντός πέντε ημερών. Επίσης χρειαζόμαστε μία τράπεζα δεδομένων. Δεν χρειαζόμαστε μία ευρωπαϊκή αρχή η οποία θα τα πράξη, διότι τότε θα τρελαθεί και συμφωνούμε όλοι ε, ότι ε, επαγγελματικά υπάρχει ε, ένα ενιαίο επίπεδο αλλά αν ο καθένας ρυθμίζει τα του οίκου του στη χώρα του τότε τίποτα δεν θα μπορέσει να προχωρήσει. Υπάρχουν και ορισμένα προβλήματα και αυτό τόσο μεταξύ ε, των πολιτικών ομάδων όσο και μέσα στην πολιτική μας ομάδα. Διότι ορισμένοι λένε εντάξει να χωρίσουμε ε, το δίκτυο από την επιχείρηση, αυτό είναι το α και το ω. Ναι μεν συμφωνούμε, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ποια θα είναι η υποδομή. Διότι υπάρχουν δίκτυα και δεν υπάρχει πρόσβαση και υπάρχουν ορισμένοι που ζητούν ε, να χωριστούν τα δίκτυα αλλά μέσα στις τροπολογίες τους ε, ε, εξαιρείται παραδείγματο χάρη το τούνελ κάτω από τη μάχη ή εξαιρείται η μεταφορά μεγάλης ταχύτητας και όσες από αυτές τις ρυθμίσεις είναι διασυνοριακές από την αρχή του 2000 δεν τις Οπότε υπάρχουν διάφορες αρχές σε όλα τα επίπεδα, διάφορες διακρίσεις τις οποίες πρέπει να αποφεύγουμε. Επίσης νομίζω ότι αυτό που δεν λειτουργεί στην πράξη ίσως με καλή πρόθεση είναι ότι πρέπει να υπάρχει ένας οργανισμός ο οποίος όμως θα προεδρεύεται από κάποιον ο οποίος θα έχει δουλέψει παραδείγματος χάρη σε σιδηροδρομική επιχείρηση για δύο χρόνια ε, όταν με ρώτησαν ποιος θα γίνει ο επόμενος ε, υπουργό μεταφορών στη Γερμανία είπα ότι δεν ήξερα ποιος θα είναι αλλά θα είναι κάποιος ο οποίος δεν έχει ασχοληθεί ποτέ στη ζωή του με μεταφορές και έτσι ήταν η τέλη, οι έξι τελευταίοι υπουργοί μεταφορών στην ε, ε, Γερμανία δεν έχουν ιδέα πώς πρέπει να προχωρήσουν και εγώ είμαι αντίθετο σε μια τέτοια λύση. Βέβαια η ρυθμιστική αρχή πρέπει να είναι ανεξάρτητη, αλλά αυτό δεν έχει, γι' αυτό δεν έχει σημασία αν υπάρξει προεργασία ή όχι διότι παραδείγματος χάρη υπάρχουν ε, περιοχές όπου δεν υπάρχει κεντρική αρχή, ε, κρατική αρχή σιδηροδρόμων και ξέρουν πώς ε, κινείται κανείς εναντίον των μονοπωλίων και εάν ένα τέτοιο άτομο με τέτοια πείρα θεωρηθεί ότι μπορεί να οριστεί σαν διευθυντής τότε πιστεύω ότι δεν θα επιτύχουμε υποχρεωτικά και αυτό ισχύει γενικά. Δηλαδή ε, νομίζω ότι θα πρέπει ε, ιδίως να υπάρξει πείρα για το τι πρέπει να διορθωθεί. Ε, λέγεται επίσης ότι θα υπάρξει μία εξαίρεση για τα κράτη της Βαλτικής αλλά και για τις τρίτες χώρες, παραδείγματο χάρη μεταξύ ε, της Ελλάδος και της Τουρκίας, ίσως γιατί οι σιδηροτροχές ε, δεν ε, συνεργάζονται, αλλά όχι μόνο εκεί. Και δεν πρέπει να αναφερόμαστε μόνο τότε στα κράτη της Βαλτικής, σαν να είναι τα μόνα όπου έχουμε προβλήματα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκρός. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που έχουν ήδη λεχθεί, αλλά θέλω να κάνω ορισμένες διευκρινήσεις. Ότι στη συζήτηση αυτή, όπως το είπε και ο κύριος Στέρξ, έχουμε κάθε συμφέρον να δώσουμε ένα σαφές μήνυμα στο Συμβούλιο από το πλευρά της Επιτροπής μας και να τους πούμε γιατί ζητούμε αυτή την αναδιατύπωση. Το είχα πει και στην προηγούμενη συνεδρίαση. Εάν ανοίξει η αγορά και όλοι έχουν ελεύθερη πρόσβαση θα αυξηθεί το ποσοστό του σιδηροδρόμου, θα υπήρχε ανάπτυξη σε όλες τις χώρες, το θέμα θα προχωρούσε ε, άμεσα ε, και θα γινόταν αυτό που δεν έγινε πριν από 10 χρόνια. Αλλά υπάρχει μία αγορά η οποία ακόμη είναι σαφώς ε, εθνική, επιχειρήσεις οι οι οποίες είναι καταχρεωμένες, ε, δεν έχουν προχωρήσει οι χώρες και δεν αυξάνεται η συμμετοχή στα ποσοστά της αγοράς. Υπάρχουν ε, ορισμένες καλές εξαιρέσεις όπου υπάρχει μία ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή. Δεν θέλω να προχωρήσω μέχρι του σημείου όπου θα πω ότι πρέπει αυτός ε, ο διευθυντής να έχει προεργασία στους σιδηροδρόμους δηλαδή ε, μπορεί να γίνει κανείς ε, δασοκόμος χωρίς υποχρεωτικά να ε, έχει εργαστεί στα δάση προηγουμένως αλλά θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος και στη λήψη αποφάσεών του και στη χρηματοδότησή του και από επιχειρήσεις πράγμα το οποίο ισχύει σε ορισμένα κράτη. Αν πετύχουμε κάτι τέτοιο τότε θα προχωρήσουμε. Αν υπάρχει προσωπικό το οποίο είναι σωστά εκπαιδευμένο εκπαιδευμένο και αμείβεται σωστά θα προχωρήσουμε, ε, θα πρέπει όμως ε, να κάνει μελέτες. Δεν ε, πρέπει απλώς να νομίζουμε ότι ο ρυθμιστής θα τα ξέρει όλα. Καλό είναι να μπορεί να προχωρήσει για να είναι και αποδοτικός. Ε, αν θέλουμε ε, να συμβάλλουμε και στην επίλυση των προβλημάτων πρέπει ε, να δούμε ότι ένα από τα μεγάλα εμπόδια που είναι η αδειοδότηση από τη μία χώρα στην άλλη θα μπορούσε να ανατεθεί εις τον ρυθμιστή για να το προωθήσει Εις, ε, όσον αφορά τις ε, υποδομές ε, και τη χρηματοδότησή τους το θέμα έχει προχωρήσει. Θα πρέπει λοιπόν το άτομο το οποίο θα αναλάβει αυτό το έργο να έχει κατευθυντήριες γραμμές. έχει δίκο και ο κύριε Στέρκ γι' αυτό. Δεν είναι δυνατόν ορισμένα έξοδα να μην συνυπολογίζονται και μετά κανείς να μην είναι υπεύθυνο για αυτές τις δαπάνες. Γι' αυτό και χρειάζεται ένας διοικητής για τις υποδομές, να υπάρχει σωστή χρηματοδότηση και να μην ξεχάσουμε τις συζητήσεις που έχουμε κάνει στο παρελθόν. Διότι ε, ε, και εγώ πιστεύω δεν πρέπει να μιλήσουμε μόνο για τα κράτη της Βαλτιστής αλλά υπάρχουν χώρες οι οποίες συνεργάζονται με τρίτες χώρες οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη αλλά και μικρές χώρες όχι μόνο το Βέλγιο αλλά και το Λουξεμβούργο θα πρέπει ίσως να μην υπάρχουν ακριβώς εξαιρέσεις αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το μέγεθός τους δηλαδή και αυτές θα πρέπει να έχουν έναν ισχυρό ρυθμιστή και θα βοηθήσει και τις μικρές χώρες να προωθήσουν το σιδηροδρομικό έργο πιο και τέλος, εάν θέλουμε να απαντήσουμε ναι ή όχι στην αναδιατύπωση, αυτό που δεν θέλουμε είναι να έχουμε δύο μεγάλες επιχειρήσεις στο μέλλον στην Ευρώπη, μία για τις εμπορευματικές μεταφορές και μία για τους επιβάτες και ε, δεν θέλουμε να φύγουμε από το κρατικό μονοπόλιο επιπλέον για να βρεθούμε σε δύο ιδιωτικά μονοπόλια. Πρέπει λοιπόν να ετοιμάσουμε το έδαφος για να μπορέσουν να επιβιώσουν οι μικροί, να υπάρχει πρόσβαση στην αγορά και εγώ προτείνω το θέμα αυτό να κλείσει διότι δεν ε, ε, είναι σωστό να λέει κανείς ότι εγώ δεν είμαι υπέρ του unbundling αλλά θέλω τόσα πράγματα που είναι unbundling κατά βάθος στην Επιτροπή θα πρέπει να ψηφίσουμε υπέρ ή κατά των δύο θεμάτων και μετά να θέσουμε το τελικό ερώτημα θέλουμε unbundling ή όχι για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε ε, για να μπορέσει να επιληθεί το θέμα αυτού του φακέλου και δεν θέλω να συζητάμε ε, SAE αν το unbundling είναι καλύτερο ή όχι πρέπει στο τέλος να ξέρουμε ακριβώς τι θέλουμε και πώς θα το εφαρμόσουμε εφαρμόσουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και όσους συνεργάζονται μαζί της για τις προσπάθειες που καταβάλουν ε, ούτως ώστε να εξευρεθεί λύση. Γιατί πραγματικά μιλάμε για τη λειτουργία της αγοράς και για την δημιουργία ισότιμων όρων για τους ε, φορείς εκμετάλλευσης. Θα ήθελα όμως να μιλήσουμε και για πιο αποτελεσματικούς σιδηροδρόμους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε επίσης ε, τον αντίκτυπο της τεχνικής διαλειτουργικότητας, κάτι το οποίο λείπει. Βέβαια, ο στόχος και το αντικείμενο αυτού του θέματος δεν είναι η διαλειτουργικότητα, η τεχνική διαλειτουργικότητα, πάντως αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις μεθόδους εργασίας, υπήρξαν κάποιες, ε, κάποιοι δισταγμοί από πλευράς εισηγητών, αλλά τώρα νομίζω είμαστε στο σωστό δρόμο. Ο καθένας ε, κάπως ε, έχει αποκρισταλώσει τις απόψεις του. Βέβαια, δεν θα συμφωνήσουμε εντελώς σε σχέση με κάποιες προκλήσεις, με κάποια πράγματα τα οποία διακυβεύονται. Η εισηγήτρια μας μίλησε για τη ρυθμιστική αρχή. Νομίζω ότι είμαστε κοντά στη συμφωνία. Σε ό,τι αφορά επίση τη χρηματοδότηση των διαχειριστών υποδομών και τη κατεξουσιοδότηση πράξη, επίση κάπω ε, τα βρίσκουμε. Σε ό,τι αφορά τώρα τη διαφάνεια, νομίζω ότι εκεί επίση θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε συνένεση. Συμφωνώ με τον Ματιέ στο ότι μετά θα πρέπει να συζητήσουμε για τις δομές Έχουμε τη σύνδεση, την αποσύνδεση, το bundling και το unbundling. Ας ολοκληρώσουμε τα άλλα και ερχόμαστε και στις δομές. Ακούγοντας τους ε, συναδέλφους, να πω πρώτα απ' όλα ότι συμφωνώ μαζί του όταν διαρωτάται για το ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πράγματι, ενίοτε τίνουμε να περιπλέκουμε τη ζωή μας και τα πράγματα. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψη της ε, Κομισιόν. Πιστεύετε ότι θα έπρεπε αυτόματα να αποφαίνεται πάνω σε οποιαδήποτε πρόταση ή απόφαση λαμβάνουν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές ή θεωρεί ότι θα έπρεπε να είναι ένα είδος ε, φορέα προσφυγής. Θα πρέπει να το σκεφτούμε λίγο περισσότερο αυτό το ζήτημα του αυτόματου χαρακτήρα. Τώρα, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να ενισχυθούν. Θα πρέπει να προετοιμάσουμε επίσης το έδαφος για μια ευρωπαϊκή η ρυθμιστική αρχή. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε με το στόχο αυτό. Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση του διαχειριστή υποδομών, θέλω να πω ότι πράγματι όταν εκπονούμε μια στρατηγική είναι φυσικό να ερχόμαστε σε διαβουλεύσεις και συνεννοήσεις με πολλούς. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας στο τέλος το αποτέλεσμα όλων αυτών των διαβουλεύσεων. Δεν είναι κακό πάντως. Παραδείγματο χάρη οι χρήστες να πούν την άποψή του. Μου φαίνεται λογικό. Τώρα, κατά πόσο αυτό πρέπει να αναφέρεται ρητά, αλλά θεωρώ ότι είναι λογικό να ακούμε τον χρήστη και γιατί όχι να το γράψουμε ότι πρέπει να τον ακούμε τον χρήστη. Πάντω ο διαχειριστής να θα λάβει την τελική απόφαση. Ένα πιο γενικό σχόλιο, το είπαν και άλλοι προλαλήσατε. θα πρέπει να μα απασχολήσει ο βαθμό λεπτομέρεια όλων αυτών των διατάξεων. Ήδη έχουμε πει πολλά, αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα για τα οποία θα πρέπει να γίνει λόγο. Και εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να είναι όσο το πιο απλό το όλο θέμα. Και τελικά ο στόχος μας θα πρέπει να είναι να υπάρχει συνέπεια, συνεκτικότητα. Σε ό,τι αφορά τη μέθοδο λοιπόν, θέλω να πω ότι ακόμη και αν συμφωνούμε για κάποια μερικά ζητήματα, τελικά νομίζω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε το σύνολο για να δούμε την γενική, την συνολική συνεκτικότητα του σχεδίου και δεν πρέπει να χάσουμε από το μυαλό μας ποιο είναι ο στόχος μας. Στο τέλος θα έχουμε και αποτελεσματικού σιδηροδρόμου, θα έχουμε και ε, πελάτες. Θα έχουμε μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα με μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς για τους σιδηροδρόμους. Υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία ακόμη δεν έχουν θυγεί και θα ήθελα είτε στις ε, συμβαστικές προτάσεις που επιπλέον στον Ρωμέλη, είτε στη συζήτηση να αναφερθούν, επί παραδείγματι η επικοινωνία σε περίπτωση κρίσης. Στο Βέλγιο αλλά και σε άλλες χώρες ενίοτε υπάρχουν κάποια ατυχήματα, συνδρομικά ατυχήματα. Το πρόβλημα είναι ότι ο φορέα εκμετάλλευση εξαρτάται από το διαχειριστή της υποδομής και μέσω πολλών άλλων ενημερώνεται για το πρόβλημα. Και υπάρχει πρόβλημα επικοινωνία, η οποία ε, κακή αυτή η επικοινωνία οδηγεί σε καθυστερήσεις. Θα έπρεπε να είμαστε πολύ πιο έτοιμοι να αντιδράσουμε, ιδίως σε περίοδους κρίσης. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους καταναλωτές και τους πελάτες, τους επιβάτες, θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες ε, πολύ εύκολα. Έχουμε το iPad, το iPhone σήμερα, όλες αυτές τις τεχνολογίες, τις εφαρμογές που μπορεί κανείς να τις μεταφορτώσει για να δει τα ωράρια των αεροπλάνων, παραδείγματος χάρη. Για τις σιδηροδρόμους δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. με ένα πάτημα του ποντικού του υπολογιστή ή ε, με το πάτημα ενός ε, πλήκτρου του iPhone να μπορεί κανείς ε, να ξέρει τα ωραία του στον δρόμο, στο Βέλγιο, στην Ισπανία. Αυτό θα διευκόλυνε πιστεύω τους επιβάτες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα, δεν θα επαναλάβω αυτά που ήδη ελέγχνησαν, αλλά θέλω να σας πω ότι πιστεύω ότι πρέπει να συγχαρούμε την υπεύθυνη ότι προχωράμε σε ένα δύσκολο δρόμο διότι η κατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου δεν είναι καθόλου ικανοποιητική στην Ευρώπη και αυτό το οποίο μιλάμε για τις πράσινες βιομηχανίες δεν θα εφαρμοστούν εάν δεν έχουμε ένα αποδοτικό σιδηροδρομικό σύστημα το οποίο δεν μπορεί να συνεχίσει αγωνιστεί αυτή τη στιγμή τις οδικές μεταφορές. Υπάρχει πραγματικό πρόβλημα. Πρέπει αυτό το σύστημα να ανοίξει, να γίνει ανταγωνιστικό, να δώσουμε τις δυνατότητες στην Ευρώπη να έχουν μια εναλλακτική λύση από τις οδικές μεταφορές. Αλλά ε, είμαστε ε, στην κατάσταση αυτή 10 χρόνια μετά από το πρώτο σιδηροδρομικό πρόγραμμα επειδή τότε το πρώτο ε, πακέτο δεν εφαρμόστηκε. Δεν θέλω λοιπόν να ξεκινήσουμε πάλι με περίπλοκα θέματα ε, τα οποία μπορούν ο καθένας ε, να τα ερμηνεύσει διαφορετικά και να υπάρχουν ε, μορατόριου. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε σαφείς ως προς τις θέσεις που θα διατυπώσουμε. Δεν θέλω σήμερα να αναφερθώ στις λεπτομέρειες των τροπολογιών. Πολλά ελέγχθησαν, χρειάζεται όμως ένα ένας εθνικός ε, υπεύθυνο για το σύστημα ε, να μπορεί να κάνει τη δουλειά του υπό καλές συνθήκες, όλοι συμφωνούν σε αυτό. Θα πρέπει να υπάρξει ένας πανευρωπαϊκός έλεγχος και αυτός θα χρειαστεί όσο πιο δυνατός είναι ε, η εθνική επιχείρηση διότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να προσεγγίσουμε την αναθεώρηση του σιδηροδρομικού πακέτου με ε, το, τη δεύτερη πτυχή που είναι η ασφάλεια και η αλληλεπίδραση. Εάν αυτά δεν συνδυαστούν με την αναδιατύπωση δεν θα υπάρξει απελευθέρωση των σιδηροδρόμων. Πρέπει επίσης να υπάρξουν ε, και κανόνες απλή ε, οι οποίοι θα γίνουν αποδεκτοί τι από τα κράτη αναλόγως του μεγέθης του, της γεωγραφικής τους θέσεως, ε, της κυριαρχίας τους. Βλέπετε λοιπόν ότι η πίση και η σαφήνεια θα ε, διευκολύνουν να γίνει αποδεκτό από το Συμβούλιο. Όσον αφορά το unbundling, δηλαδή την αποδέσμευση, θα πρέπει καταρχήν να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μιλήσουμε πιο ανοιχτά. Θα πρέπει να υπάρχει ένα πολύ περίπλοκο θέμα για το καμποτάζ των διεθνών γραμμών σε εθνικό επίπεδο αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει εκεί ε, συνεχής διένεξη και αν ήμασταν απλοί θα είχαμε αποφύγει όλα αυτά τα προβλήματα. Πρέπει το όλο το σύστημα να παραμείνει απλό διότι στο τέλος λέμε ότι δεν θα αποδεσμεύσουμε τελείως αλλά θα, υπάρχει ε, τόσο, θα υπάρχουν τόσοι περιορισμοί που δεν μπορούν καν να χαιρετηθούν και να σφίξουν τα χέρια τους ας συνενθούν στο δρόμο. Λοιπόν, ε, ε, όσο θα, πιο απλοί θα είμαστε, όσο πιο σαφείς θα είμαστε και όσο περισσότερο θα εξασφαλίσουμε την ασφάλεια και την αλληλεπίδραση τότε θα περισσότερο θα δώσουμε εις ε, το σιδηρόδρομο τη δυνατότητα να συναγωνιστεί τις οδικές μεταφορές με πράσινη προοπτική και με μέλλον. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πέρκλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ ε, θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια αλλά ε, θέλω να κάνω ορισμένες διορθώσεις πολλά ελέγχθησαν αλλά είναι βασικά θέματα νομίζω ότι για μένα είναι βασικό ε, να ξαναστρέψουμε το βλέμμα στην αρχή δηλαδή στους στόχους που επιζητούμε το είπε και ο προλαλής σας διότι πρέπει να αποβλέπουμε σε μια εναλλακτική λύση από τις οδικές μεταφορές που να επιτρέπει ελεύθερη διακίνηση στην Ευρώπη το οποίο είναι προφανές για τις αεροπορικές μεταφορές παραδείγματος χάρη για τα προγράμματα για την αγορά των εισιτηρίων να μην υπάρχουν ε, τεχνητοί φραγμοί να υπάρχει πρόσβαση στην αγορά και αν αυτός είναι ο στόχος που θα διατυπώσουμε δεν θα περιπέσουμε ή στο λάθος να προσπαθήσουμε να επισέλθουμε σε υπερβολικές ρυθμιστικές λεπτομέρειες. Είμαι νέος σε αυτή την Επιτροπή. Δεν γνωρίζω ορισμένα θέματα τόσο πολύ όσο πολύ από εσά. Αλλά όταν βλέπω ορισμένα θέματα πιστεύω ότι κινδυνεύουμε σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αν θέλουμε να κάνουμε μία τόσο λεπτομερή ρύθμιση όσο το πράττουμε στην τωρινή πρόταση ώστε το Κοινοβούλιο να είναι ο, ο ε, ε, υπέρτατος ρυθμιστής ε, και τελικά θα χάσει τον στόχο και θα μπλεχτεί στις λεπτομέρειες. Να αναφέρω ορισμένε λεπτομέρειες παραδείγματο χάρη εις ε, την δεύτερη συμβιβαστική τροπολογία δηλαδή μεταξύ του 6 και του 7 που αναφερόμαστε ει ε, τον διαχειριστή των υποδομών όπου παραπέμπουμε σε παραρτήματα για ε, μέλη του διακητικού Συμβουλίου που δεν θα μπορούν να υπερβούν μία υπηρεσία δύο ετών αλλά υπό όρους θα μπορέσουν να μείνουν τρία πάρα πολλές λεπτομέρειες ορισμένα από αυτά πρέπει να διαγραφούν διότι ακόμη και σε αυτήν την ε, συμβιβαστική πρόταση για το παράρτημα δεν πρέπει να είμαστε τόσο λεπτομερείς και αν δούμε την τροπολογία 13 θα μας επιπλήξουν ότι δεν σκεφτόμαστε επιχειρηματικά διότι πρέπει ε, να υπάρχουν υπηρεσίες που προσφέρονται ελεύθερα και αυτός ο οποίος ε, ε, δεν προσφέρει υπηρεσίες δεν πρέπει μόνο να μην χρειαστεί να δικαιολογηθεί αλλά δεν πρέπει να βρει και έναν ανταγωνιστή ο οποίος θα του διαμορφώσει κάποια τιμή θα πούμε ότι απλώς δεν προβλέπεται κάτι τέτοια ή αρνείται κάποιος ε, όλοι αυτοί οι υπολογισμοί, ε, το είχαμε συζητήσει και για τις οδικές μεταφορές, περιτεύουν. Καλό θα ήταν να μπορούμε να πούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μία ισοτιμία μεταξύ του φορτηγού αυτοκινήτου και του σιδηροδρόμου και όπου μπορεί κανείς να κάνει προσαρμογές για το κόστος του θορύβου και τα λοιπά, να μπορέσει να ε, σοφαρίσει με την κατάσταση των σιδηροδρόμων. Δηλαδή υπάρχουν διάφορα θέματα τα οποία πρέπει να υποβιβάσουμε για να αναβαθμίσουμε τα βασικά στοιχεία, δηλαδή να πούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι υπέρ αυτών των θεμάτων για την ελεύθερη πρόσβαση στις σιδηροδρομικές ε, υπηρεσίες με περισσότερη ποιότητα, διαφάνεια και ε, καλές τιμές. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και όλους τους συνεργάτες, ο κύριο Τζασάντα. Έχω κάποιες παρατηρήσεις σε σχέση με τις συμβαστικέ τροπολογίες και θέλω να φέρω δύο θέματα. Πρώτα απ' όλα την ηχορύπανση και μετά τη χρηματοδότηση. Στο παράρτημα 8.1 και στο 5. Κατά την άποψή μου, η μεθοδολογία ε, των ε, του καθορισμού των τιμών για την πρόσβαση ε, στο δίκτυο θα πρέπει να εφαρμόσετε στο πλαίσιο ενός εφαρμοστικού κανονισμού και ο διαχειριστής ε, θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του χρόνο για να εφαρμόσει προοδευτικά ε, τις διατάξεις αυτές. Ξέρουμε ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά στις μεθοδολογίε που εφαρμόζουν τα διάφορα κράτη-μέλη και δεν μα έχει δώσει η Κομισιόν μια ανάλυση που θα δείχνει πώ υπολογίζονται οι τιμέ του παραρτήματος 8. Αυτό λοιπόν το σημείο πρέπει να καταργηθεί, να διαγραφεί και η μεθοδολογία ως της πράξης θα πρέπει να βασίζεται σε εις βάθος αναλύσεις. Αυτό λείπει αυτή τη στιγμή από την πρόταση της Κομισιόν. Σε ό,τι αφορά τις ε, μειώσεις ε, τιμών, για να υπάρχει έκπτωση θα πρέπει να υπάρχει πλήρης διαλειτουργικότητα και σε ό,τι αφορά το τροχείο υλικό και σε ό,τι αφορά τις υποδομές. Η πρόταση που έχουμε αναχείρας θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια αφορές ακαμετάλλευσης, να θελήσει να εξισορροπήσει, να σταθμίσει την απώλεια κέρδου σε ένα συγκεκριμένο τμήμα, αυξάνοντας την τιμή σε μια άλλη ε, κατηγορία υπηρεσιών επειδή το κόστος των μεταφόρων και οι κοινοί κανόνες για τον καθορισμό δεν έχουν ακόμη θεσπιστεί, η προτινόμενη λύση σε ό,τι αφορά το θόρυβο είναι πρόημη, πρόορη. Στη Λευκή της Βίβλου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την εκπόνηση κοινού κανόνα για την χορύπανση και αυτό μέχρι το 2020. Νομίζω ότι το τροχαίο υλικό πρέπει να διαθέτει τους κατάλληλους μηχανισμούς, ε, τα κατάλληλα συστήματα. Και αυτό ίσως να είναι μεγαλύτερο κίνητρο από την ε, ε, τιμή. Παραδείγματος χάρη μειωμένη τιμή για όσους φορείς εκμετάλλευσης διαθέτουν πιο αποδοτικό, λιγότερο θορυβόδες, τροχαίο υλικό αυτό θα έχει ίσως αποτέλεσμα να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση στην αγορά όσοι ε, φορείς δεν έχουν αυτό το τροχαίο υλικό στη διάθεσή τους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Καντσιάν. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Σερακιάνη και όλους όσους ασχολούνται με το συγκεκριμένο έγγραφο. Σίγουρα δεν είναι εύκολο αυτό που κάνουν και δεν είναι εύκολο να βρεθεί εναρμόνιση σε κάποια ουσιαστικά σημεία. Θα ήθελα να πω το εξή. Στα όσα έχω μπροστά μου, που είναι τα συμβιβαστικά κείμενα, στη σελίδα 13 για το άνοιγμα της αγοράς, γράφει no text so far. Δεν έχουμε κείμενο μέχρι τούδε δηλαδή. Η ουσιαστική σελίδα κατά την άποψή μου για τη συζήτηση είναι ακόμα κενή και δεν γνωρίζουμε τι συμβαίνει με τα θέματα της απελευθέρωσης της αγοράς. Ακούσαμε από πολλούς ε, να αναφέρουν το ζήτημα, αλλά η συγκεκριμένη σελίδα και το κεφάλαιο 4 δυστυχώς ακόμα δεν είναι διαθέσιμη, αν θέλετε. Το λέω αυτό διότι το θέμα της απελευθέρωσης θα πρέπει να προηγείται ρητά οποιασδήποτε άλλη ε, ρύθμισης που έχει να κάνει με τη δομή δεν μπορεί να αρχίσουμε να περιπλέκουμε μόνοι μας τη ζωή μας και να μην μπορούμε στη συνέχεια να έχουμε πρόσβαση στην ελεύθερη αγορά. Δεν λειτουργούν έτσι τα πράγματα. Εγώ θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω εάν υπάρχει δυνατότητα να πάμε σε απελευθέρωση της αγοράς ή όχι. Για μένα αυτό είναι το σιώδες ερώτημα. Ο ρυθμιστής είναι ισχυρός και σημαντικός αν είναι ελεύθερη η αγορά. Ο διαχωρισμός είναι σημαντικός, το unbundling δηλαδή, και μπορούμε να φτάσουμε ε, μέχρι το τέλος εάν μπορέσουν αυτές οι δομές να λειτουργούν ελεύθερα στην αγορά και νομίζω ότι αυτό λοιπόν είναι το ουσιαστικό ζήτημα της συζήτησης. Το άλλο ζήτημα που με απασχολεί είναι το λεγόμενο τελευταίο χιλιόμετρο το αποκαλώ εγώ και εδώ. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να είμαι παραγωγική με τους τροχούς και δεν μπορούμε να είμαι παραγωγική και με οποιαδήποτε άλλη δομή μεταφοράς εάν δεν μπορούμε να διασυνδέσουμε πρακτικά και απλά τις ροές με τους μεγάλους κόμβους. Αυτές είναι οι δύο βασικές προϋποθέσεις. Όσον αφορά το διαχωρισμό λοιπόν των υπηρεσιών, ε, Καταρχάς υπάρχει το στοιχείο ότι πρόκειται για δύο πολύ σημαντικέ δομάς, γιατί υπάρχει η διοκτησία της υποδομής και η διαχείριση της αφετέρου, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να κυλούν τα τρένα στις σιδηροτροχέ και να ε, τρέχουν και τα τρένα. Πρόκειται λοιπόν για δύο βασικές αυτόνομες ε, υπηρεσίες, αλλά επειδή εδώ υπάρχει ανάγκη να καταλήξουμε σε συμβιβασμό, θα έπρεπε μέσω αυτής της σελίδα η οποία μας προτάθηκε να ε, κάνω κάποιες ερωτήσεις και να προσπαθήσω να κατανοήσω τα εξής. Στο σημείο ε του παραρτήματος για το unbundling, ποιος είναι αυτός ο οποίος ε, διορίζει το διαχειριστή του συστήματος, ποιος είναι αυτός που υλοποιεί το επιχειρηματικό σχέδιο της επιχείρησης και βάσει αυτών νομίζω ότι στη συνέχεια θα μπορέσουμε να δώσουμε μια απάντηση προκειμένου να ορίσουμε και αυτό το συμβιβασμό μεταξύ των δύο ε, αυτών επιχειρήσεων που κατ' εμέ θα πρέπει να είναι ξεχωριστές αλλά θα πρέπει να καταλήξουμε και στο σχετικό συμβιβασμό. Υπάρχουν και κάποια σφάλματα που έχουν να κάνουν και με τη δομή και τη σύνταξη. Θα έπρεπε ίσως η Γραμματεία να τα διευκρινίσει και να τα ε, εξηγήσει διότι αναφέρομαι και εγώ εδώ και υπάρχουν και κάποιες παραπομπές σε πράγματα τα οποία δεν είπα και δεν έχω θέση. Δύο-τρία πιο τεχνικής φέσεως ε, θέματα θα μπορούσα ίσως να τα κάνω και με ε, την εισηγήτρια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να κάνω και εγώ κάποια σχόλια. Είναι ενδιαφέρον να κάθεται κανείς εδώ ψηλά και να ακούει τι έχουν να πούν οι βουλευτέ. Πρόεδρευσα και το συνεδρίαση των σκιωδών στο Στρασβούργο τον Ιούλιο. Η στάση που βλέπω τώρα να διαγράφεται δεν ήταν αυτή η οποία είχε προκύψει από τη συνεδρίαση των συντονιστών, των σκιωδών μάλλον, όπου εκεί είχαμε προβλήματα και προβλήματα και προβλήματα. Κάποιοι λέγανε πρέπει να μείνει απλό και ας προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία. Άρα από κάποιες πλευρές συμφωνώ. Καλό θα ήταν ίσως ε, στη συνεδρίαση των σκιωδών εισηγητών να είχε έρθει όλη η ομάδα, η Επιτροπή μας. Έτσι θα είχαμε λύσει κάποια προβλήματα. Γιατί ποια είναι η ουσία, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι οδυνηρά αργή όλη η διαδικασία. Και θα πρέπει να έχουμε υπόψη ποιε είναι οι υποχρεώσεις μας. Μέχρι τον Νοέμβριο πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει τη θέση μας. Το Συμβούλιο ήδη έχει θέση και με τους ρυθμούς που ε, κινούμαστε είναι η ταχύτητα του μουτζούρι και όχι του τρένου υψηλής ταχύτητας. Πρέπει να επιταχύνουμε λίγο. Και πρέπει να σκεφτούμε γιατί το κάνουμε αυτό, ποιο είναι το ενδιαφέρον που έχουμε. Γιατί πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα. Γιατί. Γιατί στο παρελθόν έχει γίνει τίποτα. Το πρώτο συνδρομικό πακέτο που πολύ σωστά είπε ο Μίκαλ Κράμερ. Εννιά χρόνια μετά τίποτα και εξακολουθούν να γίνονται τα ίδια με τον ίδιο τρόπο, όπως παλιά. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να έχουμε υπόψη ποιες, εδώ, ποιες είναι οι υποχρεώσεις μας εδώ σε Επιτροπή και οι σκιώδεις εισηγητές και ο, οι εισηγήτρες θα πρέπει να λάβουν τις ευθύνε τους. Να δουν σοβαρά το θέμα. Είναι τεχνικό. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι άκρο τεχνική και ίσως εκεί να έγκυται και το πρόβλημα. Ίσως θέλουμε μια πιο απλή πρόταση, πιο προσταγμένη πρόταση από την Κομισιόν. Και όχι αυτό το παχύ τεχνικό εγχειρίδιο το οποίο ουσιαστικά φαίνεται να μας έχει υποβάλει. Δεν θέλω βέβαια να υπάρχει υπερρύθμιση. Αυτό που θέλω πάντως είναι ανεξάρτητοι ρυθμιστές που θα κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Θέλω τους ρυθμιστές να ρυθμίζουν, θέλω τους χειριστές των τρένων να οδηγούν τα τρένα και θέλω τους χειριστές υποδομών να διαχειρίζονται τις υποδομές. Αυτό που δεν θέλω και που μάλλον κινδυνεύουμε να έχουμε τελικά όμως είναι τους χειριστές που αναλαμβάνουν το ρυθμιστικό ρόλο, τους ρυθμιστές προσπαθούν ε, να διαχειρίζονται τις υποδομές και τους διαχειριστές των υποδομών που οδηγούν τα τρένα. Και αυτή βέβαια είναι συνταγή <clears throat> καταστροφής και αποτυχίας. Προς εκεί οδεύουμε όμως. Αργότερα ε, θα συζητήσουμε με τους Κιώδη σήμερα. Ο κύριος Κάντσιαν πολύ σωστά είπε ότι υπάρχουν σημαντικά ζητήματα από των οποίων ακόμη δεν έχουν συμβαστικές τροπολογίες. Να σου πω, Αντώνη, ότι χρειάστηκε μια ώρα για να καταλήξουμε σε συμβασμό σε έναν από τους 7 ή 8 τομείς για να καταλάβεις πόσο δύσκολη είναι η δουλειά που πρέπει να φέρουμε σε πέρας και πρέπει να υπάρχει καλή θέληση από όλου. Όλοι πρέπει να μετακινηθούμε λίγο για να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε συμβιβασμό και ίσως τελικά ε, μπορεί να προσπαθούμε να πετύχουμε το ανέφικτο. Το να στηρίξουν όλες οι πολιτικές ομάδες συμβιβασμούς που τελικά μπορεί να είναι ένα όνειρο θερμής νυχτός. Μπορεί τελικά η Επιτροπή μας να χρειαστεί να ψηφίσει ό,τι ήθελε προκύψει. Ο κύριος Ρόιτα από την Επιτροπή έχει το λόγο. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, όπως και ο Πρόεδρος είπε, πραγματικά με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η σημερινή συζήτηση. Νομίζω ότι ήταν μια συζήτηση που έβλεπε μπροστά στο μέλλον και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω κάποια σημαντικά στοιχεία και κάποιες σημαντικές ημερομηνίε ε, στο συγκεκριμένο πλαίσιο. η Επίτροπη και εγώ ως Γενικός Διευθυντής ε, πιεστήκαμε από πλευρά σας για να κάνουμε πρόταση για την αναδιατύπωση. Τελικώς στις 17 Σεπτεμβρίου πέρσι παρουσιάσαμε την πρόταση εκ παραλίλου και με διαδικασίες επιπαραβάση. Εγώ ήρθα εδώ στην Επιτροπή σας 10 ε, μέρες αργότερα για να σας παρουσιάσω την αναδιατύπωση και πλέον στο Συμβούλιο υπάρχει μια γενική προσέγγιση για την αναδιατύπωση εννέα μήνες πλέον μετά από την ε, πρόταση. Υπάρχει μια αίσθηση κατεπήγοντος την οποία εσείς την επιβάλλατε κατεπήγον υπό την έννοια ότι θα πρέπει να προχωρήσει αυτή η αναδιατύπωση ε, και ο σχετικός κανονισμός. Επί τούτου επικεντρωθήκαμε σε τρία βασικά στοιχεία. Καταρχάς η μακροπρόθεσμη στρατηγική για τις υποδομές, ε, χρηματοδότηση, όλα τα θέματα του ζυγίου πληρονόμων και τις αρχές που θα πρέπει να τα διέπουν όλα αυτά. Δεύτερον, ενίσχυση της ρυθμιστικής λειτουργίας. Και το τρίτο θέμα ήταν οι ε, ε, συμπληρωματικές υπηρεσίες ή όπως έλεγε και ο κύριος Καντσάνο αυτό το τελευταίο χιλιόμετρο. Υπάρχει το θέμα της ε, παροχής ενέργειας και ούτω καθεξής. Αυτά ήταν τα τρία στοιχεία λοιπόν στα οποία επικεντρωθήκαμε στην αναδιατύπωση αυτή και διαπίστωσα ότι υπάρχουν πάρα πολλές τροπολογίες στην έκθεση της κυρίας Σερακιάνη και στην έκθεση των σκιωδών εισηγητών. Υπάρχουν και συμβιβαστικές τροπολογίες οι οποίες οδεύουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα είμαι όμως απόλυτα ειλικρινής μαζί σας και όμως μας ανησυχούν κάποια πράγματα τα οποία είδαμε αυτή τη στιγμή. Εντάξει, είναι ακόμα υπομορφή σχεδίου, αλλά μας ανησυχούν. Να ξεκινήσω με το unbundling, ο διαχωρισμός αυτός. Όταν ήρθα στην Επιτροπή σας στις 17 ε, Σεπτεμβρίου, με ρωτήσατε τι γίνεται με το διαχωρισμό των υπηρεσιών. Και εγώ σας είπα τότε σαφώς ότι υπάρχει μια στρατηγική Στόχος μας είναι να προσφύγουμε στο δικαστήριο, να δούμε κατά πόσο το παράρτημα 5 της διάσημης αυτής ανακοίνωσης του 2006 είναι η σωστή βάση και δεν ασχολούμαστε με το θέμα του unbundling στην αναδιατύπωση την γενική προσέγγιση και την προσέγγιση που ακολούθησαν τα κράτη-μέλη αντισταθήκαμε για να μην επιστρέψουμε σε στοιχεία που είχαμε στην πρώτη δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους του 2001, αλλά η συμφωνία είναι επίσης ότι θα αφήσουμε το δικαστήριο να αποφασίσει επί των θεμάτων αυτών. και δεν θα προσπαθήσουμε εμείς στο περιθώριο να προσπαθήσουμε να ε, διορθώσουμε από εδώ και από εκεί δύο-τρία πράγματα. Δεν είμαστε υπέρ λοιπόν της χρήσης της παρούσας διαδικασίας αναδιατύπωσης για να αντιμετωπίσουμε το θέμα των bundling. Ο Αντιπρόεδρος Επιτροπής, ο Επίτροπος Κάλλας, δεσμεύτηκε να παρουσιάσει πρόταση το 2012 και την εκπονούμε αυτή τη στιγμή και αν έχει ολοκληρωθεί η αναδιατύπωση τόσο πιο γρήγορα θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε με την ε, πρόταση. Έχουμε και αξιολογήσεις αντικτύπου και γίνεται και αρκετή δουλειά και έχουμε την ε, ε, πρόταση αυτή στα σκαριά. Και υπάρχει και η πρόταση που ανέφερε ο κύριος Καντσιάν. Το θέμα της απελευθέρωσης των εσωτερικών ε, μεταφορών επιβατών. Και τα δύο θέματα αποσχολούν τους, ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα δύο θέματα αναφέρονται στη Λευκή Βίβλο και υπάρχει και ένα τρίτο στοιχείο που είναι σημαντικό, το θέμα της πιστοποίησης και της διαλειτουργικότητας. Αυτά όλα θα ε, παρουσιαστούν στα πλαίσια του 2012, αλλά Εάν αυτή τη στιγμή επιμολύνουμε τη συζήτηση της αναδιατύπωσης με όλα αυτά τα ζητήματα και να προσπαθήσουμε να ε, σώσουμε τον κόσμο των σιδηροδρόμων ασχολούμενοι με όλα αυτά τα θέματα, η πρόβλεψή μου είναι ότι θα υπάρξει μια πολύ μακρά διαδικασία διαπραγματεύσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά πάσα πιθανότητα θα κάνει μια πρόταση ε, στη διάρκεια της θητείας του Κοινοβουλίου, αλλά μπορεί και στις αρχές του 2013 ε, ή 2014 και θα έχουμε χάσει πάλι 3-4 χρόνια. Ήθελα να την κάνω αυτή τη δήλωση εδώ για το θέμα του διαχωρισμού και την απελευθέρωση των αγορών. Να περάσω τώρα σε κάποιες ε, συμβαστικές τροπολογίες. Καταρχάς, να πω ότι σε πολλές από τις συμβαστικές τροπολογίες υπάρχει μία ενίσχυση της αντίθεσης και της σχέσης που έχει η γενικότερη προσέγγιση που ακολουθείται στο Συμβούλιο, είτε αυτό αφορά την ανάπτυξη της υποδομής, ε, τους συγκεκριμένους ορισμούς, ε, της πρόσβασης ε, στις υπηρεσίες ή την ενίσχυση του ρυθμιστή. αλλά μας ανησυχούν επίσης και κάποιες συγκεκριμένες τροπολογίες όπου έχουμε την αίσθηση ότι οπισθοδρομούμε και σε σχέση με τη γενική προσέγγιση αλλά και σε σχέση με αυτά που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάποιες ε, τροπολογίες φαίνεται να εξασθενούν το κείμενο και ακούγοντας και τη σημερινή σας συζήτηση πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω. Τρία παραδείγματα θα σας δώσω. Εξισορρόπηση των λογαριασμών του διαχειριστή των υποδομών. Είπαμε ότι αυτό θα πρέπει να γίνει μέσα σε τρία χρόνια. Αυτή είναι η πρώτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Συμβούλιο δεν ήθελε τα τρία χρόνια, αλλά τουλάχιστον τα έχει συσχετίσει με τη διάρκεια των πολιετών συμβάσεων. Η δική σας συμβαστική τροπολογία δεν προβλέπει κανένα χρονικό περιθώριο. Δεύτερο παράδειγμα. Διαχειριστής ε, των υπηρεσιών. Εμείς ως Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή ζητήσαμε να υπάρχει νομικός διαχωρισμός. Αυτό είναι το τελευταίο χιλιόμετρο. Το Συμβούλιο δεν ήθελε να ακολουθήσει τη συγκεκριμένη άκουσα, αλλά ήταν διατεθειμένο να το ε, αντικαταστήσει με λογιστικό διαχωρισμό τουλάχιστον, ώστε να υπάρχει διαφάνεια, ενώ εσείς φαίνεται να θέλετε να διαχωρίσετε όλα τα ζητήματα, όλες τις απαιτήσει ε, του διαχωρισμού. Τρίτο παράδειγμα, εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Εσείς θέλετε να περιορίσετε τις εξουσίες των εθνικών ρυθμιστικών αρχών μόνο σε περιπτώσεις διάκρισης. Στην πράξη όμως υπάρχουν πολλές άλλες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα υπορβολικές χρεώσεις, ε, ακατάλληλα προγράμματα απόδοσης, ε, ακατάλληλες πληροφορίες ε, για προγράμματα συντήρησης, τα οποία θα μπορούσε να εξετάζει ο ρυθμιστής. Δεν ε, είναι θέμα διάκρισης, διότι αφορούν όλες τις ρυθμιστικές αρχές, αλλά, όλους τους διαχειριστές, συγγνώμη, αλλά εσείς δεν θέλετε να προχωρήσετε προς αυτή την κατεύθυνση. Θα μπορούσα να αναφέρω και άλλα, αλλά είναι πιο ενδιαλοχή, όπως για παράδειγμα οι κανόνες για τη χρέωση των υποδομών ή ο ρόλος που θέλετε να έχουν πράξει κατά εξουσιοδότηση. Αλλά θα ήθελα απλώς να συνειδητοποιήσετε ότι σε κάποιες από τις συμβαστικές τροπολογίες φαίνεται να οπισθοδρομούμε και ως προς τη γενική προσέγγιση αλλά και ως προς την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είμαστε υπέρ της απλούστευσης και της λιγότερης γραφειοκρατίας. Με χαροποιεί λοιπόν, να, όπως έλεγε και ο κύριος Στέρτς, ότι δεν θέλουμε να αποτανθούν σε εμάς και τα 27 κράτη-μέλη. Ήδη στους κανόνες, στο άρθρο 63, υπάρχει μια διάταξη που επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρέμβει. με κάποιο βαθμό να μην ε, επιβαρύνουμε ε, υπερβολικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με πολλές γραφειοκρατικές δομές, να μην πρέπει να ε, γίνουν όλα σε όλες τις γλώσσες. Δεν μπορεί να γίνουν αυτά σε δύο εβδομάδες ούτως ή άλλως. Επίσης, είμαστε και της άποψης ότι κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις όπως το θέμα των βαλτικών χωρών πρέπει να αντιμετωπιστεί, αλλά από τη διεύρυνση εγώ έχω μάθει το εξής μάθημα. Καμία παρέκκληση. Μπορεί να υπάρχουν μεταβατικές περίοδοι, μπορεί να υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες, αλλά μην δημιουργήσετε μια παρέκκληση χωρίς νόημα. Σε καμία περίπτωση μόνιμες παρεκκλήσεις και θα ήθελα να πω και κάποια πράγματα για κάποιε από τις παρατηρήσεις σα, αλλά δεν έχω αρκετό χρόνο νομίζω στη διάθεσή μου. Θα ήθελα να σας επισημάνω ότι όλοι έχουμε τους σιδηροδρόμους στο επίκεντρο των πολιτικών μας για τα επόμενα χρόνια. Γνωρίζουμε ότι αν θέλουμε να επιτύχουμε τους στόχους της Λευκής Βίβλου πρέπει να προχωρήσουμε. Ο Αντιπρόεδρος ε, Κάλλας ε, ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για αυτό το ζήτημα το γνωρίζετε, έχει προχωρήσει, έχει ένα συγκεκριμένο τμήμα που ασχολείται για ένα κοινό σιδηροδρομικό χώρο, αλλά να μην ξεχνάτε ότι η αναδιοτύπωση είναι μόνο το πρώτο βήμα. Θα πρέπει να δούμε και τι γίνεται με τη διαλειτουργικότητα των υλικών, τη γνωριγορότερη επιστοποίηση, την απελευθέρωση των, εσωτερικών, των εγχωρίων επιβατών, ε, το Connecting Europe, το οποίο ελπίζω να μπορέσουμε να συζητήσουμε πολύ σύντομα εδώ στην Επιτροπή σας και φυσικά και το θέμα του unbundling. Αλλά μην τα ανακατεύουμε όλα στο ίδιο καζάνι, διότι θα οδηγηθούμε σε παράλυση. Ίσως ε, δεν έπρεπε να ε, προχωρήσω τόσο πολύ, αλλά ήθελα να σας δείξω λίγο πώς έχει κατάσταση αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η κυρία Σαρακιάνη έχει το λόγο τελικά για να ολοκληρώσει και να καταλήξει. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Διερωτώ με αν ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιλούν με τόση σαφήνεια όπως μας μίλησε σήμερα ο Γενικός Διευθυντής, διότι εδώ στην αίθουσα άκουσα τον Επίτροπο Κάλλαν να λέει ότι είναι υπέρ του διαχωρισμού και να λέει ότι είναι υπέρ και μια συζήτηση για το unbundling ε, και στα πλαίσια της αναδιατύπωσης. Το έχω ακούσει επανειλημμένως και σε διμερείς ε, συναντήσεις και έχω ακούσει και άλλους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μιλούν για το ζήτημα προς αυτή την κατεύθυνση μιλάτε μεταξύ σας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι έχω την εντύπωση ότι δεν ήταν επαρκώς σαφή τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή ε, πιέζεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ε, δεν ξέρω κατά πόσον ε, θα πρέπει να το σκεφτούμε και αυτό, διότι η αναδιατύπωση μας δόθηκε με αρκετή καθυστέρηση. Τώρα μαθαίνουμε ότι υπάρχει διάθεση από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιταχύνουν τα χρονοδιαγράμματα ε, και θέλετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να περιμένει την απόφαση του δικαστηρίου και να κάνει την διατύπωση το συντομότερο δυνατόν για να προχωρήσουν οι εργασίες που έχει παρουσιάσει ο Επίτροπος. Τα μαθαίνουμε με μια κάποια καθυστέρηση αυτά. Θα ήθελα να υπήρχε μεγαλύτερη σαφήνεια και από πλευράς Επιτρόπου εγώ νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να περιμένει γιατί έχει άλλη ε, λειτουργία, δεν ε, πρέπει να περιμένει δικαστικές αποφάσεις. Καλά κάνει το Κοινοβούλιο και είναι φιλόδοξο όταν παρουσιάζεται ένα πρόγραμμα και προβλέπει τα πάντα προκειμένου να έχουμε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό σύστημα και γι' αυτό ακριβώς θεωρώ ότι καλώ κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αναφέρεται σε όλα τα θέματα που παρουσιάσαμε στην αναδιατύπωση. Υπάρχουν κάποιες συμβιβαστικέ τροπολογίες που ε, είναι ήδη γνωστέ στη σπάση και σε αυτές τις συμβιβαστικέ τροπολογίες έχει γίνει εν μέρη συζήτηση και για κάποια από αυτά τα ζητήματα. Σαφώς είμαι και διατεθειμένη να απλουστεύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τα πράγματα και για τη ρυθμιστική αρχή να προσπαθήσουμε αν ε, ε, είναι απαραίτητο να διαγράψουμε κάποια στοιχεία που επιβαρύνουν το έργο του ρυθμιστικού φορέα αλλά υπάρχουν κάποιες προβλέψεις οι οποίες έχουν παρουσιαστεί, κάποια πράγματα, έχουν, κάποιες διατάξεις έχουν παρουσιαστεί και από τους σκιώδεις συζητητές. Κάναμε όλη αυτή τη δουλειά με πρόθεση να ε, σκεφτούμε μαζί έναν ανεξάρτητο ρυθμιστικό φορέα, ο οποίος θα είναι ισχυρός και θα είναι σε θέση με διαφάνεια να διεξάγει σημαντικά καθήκοντα τα οποία θα καθορίζονται σαφέστατα και παρουσιάζονται στις συμβαστικές τροπολογίες. Όσον αφορά τώρα την απλούστευση των δραστηριοτήτων, θα δούμε κατά πόσον υπάρχει δυνατότητα να είναι πιο απλά τα πράγματα, αλλά νομίζω ότι είναι σαφές ε, προς τα που οδεύουμε. Όσον αφορά τώρα τις χώρες της Βαλτικές, Υπάρχει μια ανοιχτή αντιπαράθεση με τον κύριο Τζίλε, ο οποίος έχει αναφέρει επανειλημμένος το ζήτημα. Εγώ δεν είμαι υπέρ μιας γενικής παρέκκλησης, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες εξαιρέσεις, οι οποίες συνάδουν και με τα όσα ε, κατέληξε το Συμβούλιο επί του θέματος. Εγώ θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να κάνει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα θα πρέπει να μπορούμε να μιλάμε για εθνικό ρυθμιστό, ε, ρυθμιστή, συγγνώμη, όπως αναφέρθηκε και στους συμβιβασμούς. Θα πρέπει να μιλάμε για μεγαλύτερη διαφάνεια και μάλιστα μιλάμε για διαφάνεια και δεν μιλάμε για bundling στις ε, ε, συμβαστικές τροπολογίες και νομίζω ότι η διαφάνεια είναι αυτή που μας ενδιαφέρει στο λογιστικό διαχωρισμό, στο, λογιστικ... στο διαχωρισμό των διοικητικών συμβουλίων, δηλαδή στοιχεία διαφάνειας που διευκρινίζουν ακόμα περισσότερο το ρόλο του καθενός εκ των φορέων που ε, συμμετέχουν στο σιδηροδρομικό σύστημα, όπως έλεγε και ο Πρόεδρος Σίμψον προηγουμένως. Όσον αφορά τώρα τα υπόλοιπα ζητήματα, νομίζω ότι για τη χρηματοδότηση έχουμε καταλήξει σε καλό συμβιβασμό και για τις πράξεις κατεξουσιοδότησης ε, νομίζω ότι είναι πλέον σαφή τα πράγματα. Το ίδιο ισχύει και για το άρθρο 13 για τις υπηρεσίες. Βεβαίως και σήμερα θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας για τα συμβαστικά κείμενα. Κατά την άποψή μου δεν νομίζω ότι μπορώ να δεχτώ αυτή τη στιγμή την πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έρχεται ε, πολύ καθυστερημένα, κατόπιν εορτής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία μου όντως ε, κλείνουμε προσωρινά μία συζήτηση η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως και ακόμη χρήζει διευκρινήσεων. Περνάμε στο επόμενο θέμα τώρα που είναι η ε, συζήτηση σχετικά με το σχέδιο προπολογισμού 2012 όσο αναφορά το θέμα μας. Ο κύριος Λιμπεράση δεν είναι εδώ, οπότε δίνω τον ε, λόγο εις ε, τον αντικαταστάτη του. Ευχαριστώ. Καταρχήν ο κύριος Λιμπεράσχη δεν μπόρεσε να συμμετάσχει και γι' αυτό μου ζήτησε να αναφέρω διάφορα θέματα ε, το Και ξέρετε προχωράει η συζήτηση του προϋπολογισμού και γνωρίζουμε την ε, θέση του Συμβουλίου για ορισμένα θέματα και αυτά πρέπει να συζητήσουμε και με ορισμένες τροπολογίες θα χρειαστεί να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα αντίβαρο. Αυτό είναι κάτι που θα συζητήσω στη συνέχεια, αλλά ξεκινώ με ένα καλό νέο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έχει αντιδράσει στις θέσεις μας σχετικά με τρία προγράμματα πιλωτικά, καταρχήν σχετικά με την πολιτιστική και βιομηχανική κληρονομιά για ε, τον τουρισμό και προσβασιμότητα για όλους και για τις πληροφορίες και κρατήσεις στις μεταφορές σε όλα τα μέσα μεταφοράς. Τα, τα τρία αυτά πιλωτικά έργα ήταν ένα θέμα που μας απασχολούσε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν σχολίασε δύο εξ αυτών για την πολιτιστική κληρονομιά και τον τουρισμό. Όσον αφορά την ε, ολοκληρωμένη έκδοση εισιτηρίων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντέδρασε θετικά, αλλά υπέβαλε και τροπολογίες για να μπορέσει να συνάδει η πρότασή μας με αυτά τα οποία ήδη συζητούνται στα πλαίσια της επιτροπολογίας. Και αυτό είναι το καλό νέο. Στη συνέχεια οι μόνιμοι αντιπρόσωποι και αυτό είναι το λιγότερο καλό νέο προτείνουν να μειώσουν ορισμένα κονδύλια και αυτό φαντάζομαι στις 22 Ιουλίου θα επιβεβαιωθεί από το Συμβούλιο. Βέβαια οι προτάσεις αυτές δεν μας πλήττουν σοβαρά διότι από 10 εκατομμύρια ευρώ στον προπολογισμό του 2012 θα έχουμε μία μείωση κατά 0,6% σε σχέση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά για τις πληρωμές η μείωση είναι πολύ πιο σοβαρή 40 ε, εκατομμύρια δηλαδή 12% Οπότε πρέπει να σκεφτούμε ε, ε, γιατί υπάρχουν αυτές οι τεράστιες διαφορές. Όσο αναφορά τα TNT, τα ολοκληρωμένα δίκτυα υπάρχει μία σημαντική μείωση ε, κατά 11,5% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφαλείας της ε, Ναυσιπλοείας ε, προτείνονται ε, ε, ε, προτείνεται επίσης μία μείωση Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να θέσουμε ορισμένα ερωτήματα. Καταρχήν χαιρετίζουμε τη στάση για τα τρία πιλωτικά έργα, αλλά πρέπει να αντισταθούμε σχετικά με τον προπολογισμό, διότι το πρόγραμμά μας προβλέπει ότι οι αριθμοί του σχεδίου προπολογισμού είναι το ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο και το Συμβούλιο προτείνει κάτι πολύ χαμηλότερο και για τις υποχρεώσεις και ακόμη περισσότερο περισσότερο για τις πληρωμές. Αυτή είναι η κατάσταση του φακέλου. Όπως σας είπα, έχουμε ακόμη ορισμένες μέρες στη διάθεσή μας για να αντιδράσουμε. Ο πρόεδρος έχει θέσει ε, σαν προθεσμία την 27η Ιουλίου για τις τροπολογίες και ελπίζω ότι εν μεταξύ όλες οι πολιτικές ομάδες θα καταλήξουν σε μια κοινή στρατηγική. Ευχαριστώ και ε, επειδή η σκιώδης σε αυτό το φάκελο πρέπει να σας πω ότι καταρχήν ο, το, φάκελος που πρότεινε ο κύριος Λιβεράτσχη είναι εξαιρετικός και τον χειρίστηκε πάρα πολύ καλά η ομάδα του ΕΛΚ παρόλο που το τέρμα στο τέλος είμαστε κάπως διαφοροποιημένοι σχετικά με τη χρήση του προϋπολογισμού δεν χρειάζεται δηλαδή να περιμένουμε περιμένουμε να επιπέσουν επάνω μας οι ράβδοι για να μας μαστιγώσουν. Πρέπει να προτρέξουμε και έχουμε καλά νέα για κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει αλλά είναι ουσιαστικά επουσιώδες σχετικά με τον προκατακτικό προϋπολογισμό τουλάχιστον οι προτάσεις της Επιτροπής μας ελήφθησαν υπόψη πράγμα το οποίο ούτως ή άλλως μπορεί να βοηθήσει τον τουρισμό που είναι σε κακή κατάσταση. Οπότε ναι μεν συμφωνούμε για τον προϋπολογισμό αλλά όχι για τη σταθεροποίηση του τουρισμού. Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις ε, με τους μόνιμους αντιπροσώπους στο Συμβούλιο, ε, ξέρουμε ότι μας μειώνουν για λογιστικούς απλούς λόγους τις πιστώσεις και 12% βέβαια ο αριθμός είναι πολύ υψηλός σε σχέση με τις λογικές προτάσεις που διατυπώσαμε. Ε, δεν μπορούμε να πούμε ότι η Επιτροπή μας έκανε ε, παράλογες επιτροπές ή ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έκανε λογικές ε, επιτροπές οι οποίες έχουν διατυπωθεί αντιθέτως και πρέπει να τονίσω ότι κάποια στιγμή όπου δημοσιονομικά εξετάζουμε τις υποδομές και την εξάρτηση ε, από περιφερειακά ταμεία το να μειώνονται τα ε, διπυρωτικά δίκτυα νομίζω ότι είναι κάτι απαράδεκτο και πάλι ε, βέβαια οι οργανισμοί είναι αυτοί οι οποίοι πλήττονται και νομίζω ότι θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας και εκεί και υπάρχει μία διαφορά ε, ε, μεταξύ την αντίληψη της Επιτροπής Μεταφορών και το Συμβούλιο διότι οι οργανισμοί αυτοί είναι ο εκτελεστικό, το εκτελεστική οργάνωση ε, είτε για το Συμβούλιο είτε ε, για το ε, Κοινοβούλιο. Να θεωρήσουμε λοιπόν ότι πρέπει όλες αυτές οι δαπάνες να επιληθούν με τον ίδιο τρόπο είναι απαράδεκτο διότι καταρχήν υπάρχει μια ολοκληρωμένη ε, ναυτιλιακή πολιτική η οποία δεν ε, στηρίζεται σε τίποτα. Δεύτερον, ε, θα χρειαστεί μία αναδιατύπωση της ναυτιλιακής πολιτικής και μειώνουν και τις, και τις χρηματοδοτήσεις. Δηλαδή υπάρχει μία πλήρη αντίφαση μεταξύ των δηλώσεων για ανάγκη ολοκληρωμένων πολιτικών, ανάγκη επενδύσεων, επενδύσονται στα πλαίσια μίας, ε, ενός ευρωπαϊκού οργανισμού και εκεί συμφωνούμε με το Συμβούλιο και μετά δημοσιονομικά ε, υπάρχει μία πολιτική διαγραφής και κριζώσεως η οποία ε, δεν ήταν αυτό το οποίο εμείς είχαμε ζητήσει. Και όπως είπε ο Σαΐντ στο τέλος, το Συμβούλιο θα υποβάλει το σχέδιό του στις 22 Ιουλίου αλλά υποθέτω ότι θα ακολουθήσει τη γραμμή του, των μονίμων αντιπροσώπων του Κορεπέρ και έχουμε ελάχιστο χρόνο για τις τροπολογίες μας αλλά θα σας υπενθυμίσω ότι πέρυσι κάναμε τις προτάσεις χωρίς να έχουμε καν ε, προτάσεις του Συμβουλίου ενώ τώρα έχουμε μια εβδομάδα γνωρίζοντας τα πράγματα για να υποβάλουμε τις προτάσεις μας. Ο κύριος Στέρξ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Αντικαθιστώ την κυρία Μάγερ, την Κιζίνα Μάγερ, η οποία είχε προβλήματα με τη μέση της και νοσηλεύεται. Που έχει πάντως διαβάσει κάποιες πληροφορίες, ε, τις οποίες με τα χαρά θα μοιραστώ με τον εισηγητή που και αυτός ε, κάποιον άλλο αντικαθιστά. Λοιπόν, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Λιμπεράτσκι για τη γνωμοδότησή του πραγματικά την τη θέση της πολιτικής μας ομάδας. Παράγραφος 6 που αφορά την ε, θαλάσσια πολιτική και παράγραφο παράγραφος 6 για την τουρισμό είναι πολύ σημαντικές. Βέβαια θα καταθέσουμε και κάποιες τροπολογίες για να επανεισαγάγουμε την αρχική πρόταση προϋπολογισμού ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θεωρούμε ότι η θέση της Κορεπέρ δεν αντικατοπτρίζει επαρκώς τη σημασία που έχει ο τουρισμός για τη Στρατηγική Ευρώπη 2020. Κεφάλαιο 6.3 για τα διευρωπαϊκά δίκτυα των τομέα μεταφορών. Είναι ένα παράδειγμα. Δεν συμφωνούμε καθόλου με την πρόταση της Κορεπέρ. και δεν ε, υπηρετούμε σε καμία περίπτωση την ε, πολιτική μεταφορών όπως θα έπρεπε να είναι σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης η ομάδα μας θα ήθελε να σχολιάσει τα πιλωτικά προγράμματα. Ο Σάιντελ Καντραουή έκανε λόγο για αυτά. Θεωρούμε και εμείς ότι είναι απαραίτητο να εξακολουθήσουμε να παρασπίζουμε τα προγράμματα αυτά. Σε ό,τι αφορά το Integrated Ticketing, αυτό το τρίτο πιλωτικό σχέδιο, θα θέλαμε να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας απαντήσει γιατί αυτό περιορίζεται σε τρεις χώρες. Γιατί δεν θα μπορούσε να είναι ευρύτερο. Αυτό είναι το τελευταίο με ερώτημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Στέρξ. Κυρία Φώστερ είναι η επόμενη ομιλήτρια που φαντάζομαι εκπροσωπεί το σκιώδη της εισηγητή. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομη κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Στρέξ μας έδωσε πράγματι ένα παράδειγμα ενός πιλωτικού προγράμματος το οποίο ε, προσπίζουν. Παράδειγμα επίσης και το ΣΕΖΑΡ ε, για τον Ευρωπαϊκό Ρανο, επίσης πολύ σημαντικό. Δεν θέλω να χαλάσω την γιορταστική ατμόσφαιρα, αλλά η συνοπτική καλή έκθεση του κ. Λιμπεράτσκι. Παρ' όλα αυτά, το μόνο που μιλάμε εδώ είναι αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης, περισσότερα χρήματα, περισσότερη χρηματοδότηση. Από πού θα τα βρούμε όλα αυτά τα χρήματα όμως. Νομίζω ότι εμείς πάντοτε είχαμε ξεκαθαρίσει την άποψή μας. Όταν έχουμε πόρους στη διάθεσή μας, πρέπει να κάνουμε μια νέα κατανομή. Αν θέλουμε να έχουμε άλλα προγράμματα, θα πρέπει να βρούμε μέσα στον υφιστάμενο προϋπολογισμό κάποια άλλα χρήματα. Εδώ μιλάμε για δεκάδες ή ε, εκατομμύρια, για δισεκατομμύρια. Δεν μπορούμε να βρούμε από το αέρα χρήματα. Ναι, πράγματι έχουμε τον τουρισμό, τα πιλωτικά προγράμματα. Το, αυτό το integrated ticketing και αν δούμε τους σιδηροδρόμους ή άλλους ε, τρόπους μεταφοράς, είναι στο συμφέρον των επιχειρήσεων να το κάνουν για να αυξήσουν ε, την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να επενδύει χρήματα σε προγράμματα ε, αντί να το κάνουν οι ίδιες επιχειρήσεις που θα έπρεπε να το κάνουν. Νομίζω ότι εμείς πρέπει να στείλουμε τα σωστά μηνύματα και να ορίσουμε τις κατευθύνσεις. Αλλά αν ε, κάποιος θέλει να κάνει κάτι για οποιοδήποτε τρόπο μεταφορών, ε, μεταφοράς θα πρέπει ε, να κινητοποιηθεί η ίδια η επιχείρηση η οποία είναι προς το συμφέρον να το κάνει. Και βέβαια υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος ανταγωνισμός στον τουρισμό. Καλό είναι να προωθήσουμε αυτό το πρόγραμμα, να έρθουν όλοι να επισκεφθούν ε, την Ευρώπη. Αλλά τι άλλο να προσθέσω, ευχαριστώ τον εισηγητή, αλλά επί της ουσίας θα χαλάσω το πάρτι λέγοντας ότι ξέρετε δεν υπάρχουν άλλα λεφτά. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε με πιο σοφό τρόπο τα ε, χρήματα που έχουμε στη διάθεσή μας. Να τα χρησιμοποιήσουμε καλύτερα. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Κράμερ έχει τώρα το λόγο. Ναι, και εγώ εκπροσωπώ την κυρία Ντουρόν η οποία βρίσκεται σε ένα ταξίδι με, με αποστολή και βλέπουμε ότι ο βιώσιμος τουρισμός περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό διότι ο προπολογισμός είναι η πολιτική σε αριθμούς. Ε, αν δούμε λοιπόν τι περιλαμβάνουν οι συνθήκες θα πρέπει να ε, εφαρμόζονται. Ε, το, το, ποσό δεν είναι πολύ υψηλό αλλά εφόσον υπάρχει ένα κεφάλαιο για τον βιώσιμο τουρισμό στον προπολογισμό πρέπει να το εφαρμόζουμε. Επίσης από το 1955 έχουμε επενδύσει 50 δισεκατομμύρια στην πυρνική ενέργεια την οποία θέλουμε να κλείσουμε αύριο το πρωί. Περάσαν 20 χρόνια δεν έχουμε προχωρήσει και υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει πάλι να ξαναεξετάσουμε και να ερευνήσουμε. Δηλαδή οι σιδηρόδρομοι δεν θα, έχουν, ε, ε, ε, δεν θα μπορέσουν να λύσουν τα προβλήματά τους αν δεν λύσουν το θέμα της συγχωρήπανσης και του θορύβου και θα χρειαστούμε ε, τα μισά χρήματα και θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Έτσι πρέπει να προχωρήσουμε την έρευνα ε, και να περιλάβουμε στην ομοθεσία ότι η συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως δεν θα αναφέρεται μόνο στις υποδομές αλλά και στην αποτελεσματικότητα. Πρέπει επίσης να ξανασκεφτούμε τα, τους τα μεγάλα προγράμματα. Διότι στην Ευρώπη υπάρχουν ε, οι διάδρομοι, τους οποίους έχουμε καταρτήσει, αλλά δεν έχουμε πει πώς θα τους ε, χρησιμοποιήσουν και εφαρμόσει τα κράτη. Ε, πάντοτε υπάρχουν μεγάλα προγράμματα και έχουμε πολλά εθνικά παραδείγματα τα οποία μπορούμε να αναφέρουμε. Παραδείγματος σαν το διάδρομο από το Ταλίν μέσω Βαρσοβίας στη Μεσόγειο, ο οποίος είναι ο διάδρομος 5 και πρέπει να αναπτυχθεί σιδηροδρομικά. Αλλά θα τέμνεται σε ορισμένα σημεία με ε, τον διάδρομο προς την Μπρατισλάβα, δηλαδή Παρίσι, Βιέννη, Μπρατισλάβα και οι ε, Αυστριακοί ε, θέλουν να συνδέσουν αυτό αυτό το διάδρομο μαζί με ένα τούνελ στο Ζέμερινγκ ε, και με άλλο ένα όπου ξέρουμε ότι ε, θα είναι μία δαπανηρή ε, μεν κίνηση αλλά αντί να κάνουμε δύο παράλληλους διαδρόμους θα είναι πιο γρήγορο και λιγότερο δαπανηρό να δημιουργήσουμε ένα κοινό πρόγραμμα αντί για δύο διαδρόμους. Δεν χρειαζόμαστε υποχρεωτικά περισσότερους πόρους, αλλά χρειαζόμαστε μια ε, πιο έξυπνη πολιτική που θα διαχειριστεί καλύτερα λιγότερους πόρους. Ο κύριος Κιούν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να απευθύνω μία ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, σχετικά με το θέμα που έθιξε προηγουμένως ο κύριος Κράμερ. Δηλαδή, αν έχουμε εμπορευματικές και επιβατικές μεταφορές στο σιδηρόδρομο την επόμενη δεκαετία στην Ευρώπη με μία αύξηση κατά 10% ε, και ε, επιβαρύνουμε ιδιαιτέρως ε, τις εμπορευματικές μεταφορές η χορύπανση θα είναι πολύ σημαντική και πάντοτε ε, επενδύουμε μόνο σε υποδομές διότι έτσι προβλέπουν ε, οι συνθήκες παραδείγματος χάρη της ε, TNTS όπου είναι υποδομές και έχουμε έναν μεγάλο προϋπολογισμό ετησίως στη διάθεσή μας αλλά εις το σιδηρόδρομο και στις εγκαταστάσεις του, δεν μπορούμε να επενδύσουμε, ζητούμε να υπάρξει μία αλλαγή στο επίπεδο θορύβου, ενώ αυτό θα μπορούσε να γίνει με καλύτερα συστήματα παιδίσεως και με νέο εξοπλισμό. Αν είχαμε εξοπλίσει και προσαρμόσει ε, εγκαίρως του σιδηροδρόμους σε αυτές τις προδιαγραφές, θα είχε κοστίσει 4,5 δισεκατομμύρια εκατομμύρια θα συμμετείχαν τα κράτη-μέλη και οι σιδηροδρομικές ε, επιχειρήσεις αλλά εδώ νομίζω ότι με λίγα χρήματα θα μπορούσαμε να προωθήσουμε ένα πολύ καλό μέτρο. Ευχαριστώ. Το, ο κύριος Μπονούτσι για την ε, Επιτροπή έχει τώρα το λόγο για να απαντήσει σε ερωτήσεις αυτές. Κύριε Διευθυντά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Φυσικά η Επιτροπή στηρίζει πλήρως ε, τις προτάσεις του εισηγητή. Βέβαια έχουμε και κάποια συγκεκριμένα σημεία που πρέπει να ε, προσέξουμε. Δεν θέλω να ψέλθω τώρα σε λεπτομέρειες, αλλά θα σας ε, παρακαλέσω να δείτε πολύ προσεκτικά το όλο θέμα των οργανισμών. Είναι λεπτή η φάση. Ήδη το 2011 κάναμε προσπάθεια ε, ανάπτυξης, έκνα ανάπτυξης του προσωπικού και για το 2012 οι θέσεις που ζητούνται ή κάποιες θέσεις που ζητούνται ουσιαστικά είναι ε, το απαραίτητο για να μπορέσει οι οργανισμοί να εκπληρώσουν τα νέα καθήκοντα που ζητά το Συμβούλιο. Ιδίω ε, για την ΕΜΣΑ ξέρουμε ότι είναι τρεις οι που θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί και για την ΕΑΖΑ. Το Single European Sky ήταν το πρόγραμμα. Ε, θα πρέπει να δούμε τι πρέπει να κάνουμε με αυτές τους ε, δύο οργανισμούς και τις προτάσεις το 2012. Σε ό,τι αφορά τα άλλα θέματα που αναφέρθηκαν, έχουμε μείωση 30-32% για το Single European Sky. Άρα πρέπει να δούμε πόσο γρήγορα θέλουμε να κινηθούμε σε αυτό το τομέα. Κατά τα λοιπά νομίζω ότι η αιστεία στον τομέα της έρευνας μπορεί να γίνει με, την, ε, με τον εξορθολογισμό των στόχων μας. Και αυτό αφορά βέβαια εν μέρη και το τροχαίο υλικό. Θόρυβος, χορύπανση. Σιγά σιγά κάνουμε κάποια βήματα πρόοδου. Αν τώρα η νομική βάση πρέπει να αλλάξει ώστε να καλύψει και αυτή την ε, πτυχή, αυτό είναι κάτι το οποίο υπερβαίνει τα αμυγή δημοσιονομικά. Κατά τα λοιπά δεν έχω σχόλια να προσθέσω και πρέπει να συγχαρούμε τον εισηγητή για την ανάλυση που μας παρουσίασε. Ευχαριστώ, Πρόεδρος. Βλέπουμε ότι συμμεριζόμαστε τις ίδιες, μάλλον έχουμε τις ίδιες ανησυχίες. Δεν είναι στην αίθουσα ο εισηγητής για να του ξαναδώσω το λόγο, άρα προτείνω να περάσουμε στο επόμενο σημείο της μερισιάς διάταξης. Συγκεκριμένα πρόκειται για την έκθεση της κυρίας Λίχτενμπέργκερ που κατέφθασε. θέμα είναι η χρησιμοποίηση των προσωπικών στοιχείων επιβατών. Μιλάει βέβαια με το γείτονά της εκεί, τον κύριο Κράμερ ή βλέπω εκεί να πλέκεται ένα ειδήλιο, δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, κυρία Λίχτενμπέργκερ, είμαστε σε ένα θέμα το οποίο σας είναι προσφυλές, ίσως ε, λιγότερο από τον ε, παρακαθημένο σας, αλλά τέλος πάντων είναι το θέμα της χρησιμοποίησης των προσωπικών στοιχείων επιβατών. Πριν σας δώσω το λόγο για να κάνετε την παρουσίασή σας, να πω ότι η έκθεση του Συμβουλίου, θέλετε να τα πείτε εσείς, ε, η έκθεση του Συμβουλίου για την πρόταση του Συμβουλίου ουσιαστικά ε, θα γίνει στις 22 Ιουλίου για τον προπολογισμό. Μπορούμε να καταθέσουμε τροπολογίες μέχρι τις 27 Ιουλίου εμείς. Σε ό,τι αφορά τώρα την ψηφοφορία, η ψηφοφορία θα γίνει στις αρχές Οκτωβρίου στην Επιτροπή μας. Α, όχι, λάθος, συγγνώμη. Στις 30 Αυγούστου στην Επιτροπή μας. Μόλις έχουμε επιστρέψει ψηφιακοπές δηλαδή. 6 Οκτωβρίου στην Επιτροπή Προϋπολογισμών και στην Ολομέλεια τον Οκτώβριο. Για να μπορέσουμε πράγματι να έχουμε τη διμερή συμφωνία πριν τα τέλη του έτους. Κύριε Λίχτεμπέργκερ, ε, σας δίνω τώρα το λόγο για το PNR. Ευχαριστώ. Το θέμα των ε, στοιχείων ε, των ε, επιβατών, η, μετα... η μετάδοσή τους και η αξιοποίησή τους και στο παρελθόν υπήρξε αντικείμενο πορών συζητήσεων και αξιολογήσεων και όσοι ήταν εδώ πρόσφατα θυμούνται ότι είχαμε κάνει μία πολύ σημαντική ακρόαση με τους μυρογνώμονες του χώρου και πρόκειτο ουσιαστικά για στοιχεία από το CRS, δηλαδή από το σύστημα κρατήσεων μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και υπήρχε ότι δεν μπορούσε να διαχωρίσει κανείς τα στοιχεία κατά την χρησιμοποίησή τους και ούτω καθεξής. Στη γνωμοδότησή μου προσπάθησα ε, όλα αυτά τα οποία είχα ε, συγκεντρώσει να τα προωθήσω καθώς επίσης ε, και ε, ε, τα σχόλια της νομικής υπηρεσίας του Συμβουλίου και της αρμοδίας αρχής καθώς επίσης και τις εθνικές αποφάσεις ε, των συνταγματικών δικαστηρίων όπως στη Γερμανία παραδείγματος χάρη που επισημαίνουν ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα όσον αφορά την αναλογικότητα και την εφαρμογή και ιδίως και σχετικά με το θέμα του εάν μπορεί κανείς να επιτύχει με αυτόν τον τρόπο τον επιζητούμενο στόχο. Προσπάθησα λοιπόν σχετικά με το θέμα το οποίο μας απασχολεί ιδιαιτέρως να το προχωρήσω και πρέπει να ε, λάβουμε υπόψη το θέμα του κόστους και ε, αυτά τα οποία ε, αναφέρονται εις ε, τα θέματα της ασφαλείας καθώς επίσης και τις ασάφειες. Γι' αυτό και προσπάθησα να διατυπώσω την γνωμοδότησή μου κατά τέτοιων τρόπων ώστε οι ε, νομοθετικές αυτές εξελίξεις να ληφθούν υπόψη παρακαλώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο θέμα της ε, κατανομής των εξόδων να μας διατυπώσει ε, μία γνωμοδότηση όσον αφορά τις λεπτομέρειες στην ε, νομική απόφαση ε, διατυπώθηκε ένα πρόβλημα δηλαδή ότι είναι ασαφείς οι ορισμοί ε, τι σημαίνει σοβαρή εγκληματικότητα παραδείγματος χάνει πράγμα το οποίο οδηγεί σε μία νομική ανασφάλεια διότι εδώ μιλάμε για τη αντιτρομοκρατικά μέτρα και τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν χρησιμοποιηθούν για αντιτρομοκρατικά μέτρα και δυστυχώς αυτό ε, δεν ισχύει ε, μόνο και επίσης ε, υπάρχει ασάφεια όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων και την ε, μετάδοσή τους σε τρίτες χώρες. Αυτό είναι ένα από τα θέματα που μας απασχολεί. Όχι μόνο ε, τις ε, ανταλλαγές τις οποίες εμείς έχουμε ρυθμίσει νομικά και συμβατικά αλλά και τις περαιτέρω μεταφορές και όσον αφορά την αποθήκευση προσπάθησα επίσης να λάβω υπόψη αυτό το οποίο ελέγχθη τρόπον ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Κατά τη γνώμη μου υπάρχει ένα θέμα σχετικά με τις αεροπορικές υπηρεσίες γενικώ, δηλαδή ε, αν ε, κανείς ε, μεταβαίνει κάπου αεροπορικά δεν είναι προφανές ότι πρέπει να αποπέμψει ορασμένα συνταγματικά του δικαιώματα και ε, υπάρχει το θέμα του εμπιστευτικού χαρακτήρα και ε, της ε, μεταβίβασης των στοιχείων όπως βλέπετε εγώ προσπάθησα να λάβω υπόψη ότι υπάρχει προσυζήτηση αυτή προς στιγμή και να διατυπώσω αντιστοίχως τις τροπολογίες μου μπόρεσα να μιλήσω μιλήσω μόνο με ορισμένους από όλους τους σκιώδεις εισηγητές γιατί ε, στην ε, εβδομάδα του Στρασβούργου είχαμε πάρα πολλή δουλειά δεν μπορέσαμε να βρούμε μια κοινώς αποδεκτή στιγμή να συναντηθούμε και ελπίζω ότι έστω και διμερός θα μπορέσουμε να διευκρινίσουμε και να καταλήξουμε ε, σε συμβιβαστικές τροπολογίες, όχι βέβαια την 1η ή τη 2η Αυγούστου, αλλά διότι δεν θέλουμε, να επέμβουμε στο χώρο διακοπών των κουρασμένων ευρωβουλευτών αλλά ε, αυτή είναι η γνωμοδότησή μου σαν υπεύθυνη της ε, Επιτροπής Μεταφορών θεώρησε ότι δεν έπρεπε να αναφερθώ μόνο στην πτυχή των μεταφορών αλλά και της, νομικο... της νομιμότητος γιατί υπάρχει μία βασική αλλαγή των πολιτικών που εφαρμόζουν οι αεροπορικές εταιρείες και όταν μιλάμε για τις αεροπορικές εταιρείες αντιλαμβάνεστε ότι και αυτές έχουν ορισμένες αντιρρήσεις. Καλό θα ήταν λοιπόν να μπορέσουμε να βρούμε μία κοινή λύση στην Ευρώπη όχι όχι όπως με την κατακράτηση ε, των δεδομένων ο ένας να τα κρατάει 15 χρόνια και όλος 6 μήνους αλλά πρόκειται για νομικά θέματα και πρόκειται για στοιχεία τα οποία ε, αποσκοπούν σε ένα συγκεκριμένο ε, στόχο και γι' αυτό συγκέντρωνονται άρα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς. Ε, θα πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο αδικίας και να είμαστε πολύ σαφείς και επιμελής σε αυτό διότι δεν πρόκειται μόνο για τις αεροπορικές μεταφορές και την ασφάλειά τους αλλά και για άλλες μεταφορές και γι' αυτό πιστεύω ότι μπορεί να έχει επιπτώσεις αρνητικές γενικώ στην κινητικότητα για την, το ΕΛΚΟ κύριος Γκρός. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή ο κύριος Ντεκράν να δεν είναι εδώ και από ό,τι ξέρω δεν είχε καν χρόνο να συζητήσει μαζί σας το θέμα αυτό αλλά στα πλαίσια του ΕΛΚ θα το συζητήσουμε με τους συναδέλφους της Επιτροπής μπορώ όμως να σας πω από την αρχή ότι με την πρότασή σας προβαίνετε σε σημαντικές αλλαγές σε σχέση με το ότι έχει διατυπώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρέπει να πω ότι αν πρόκειται για την ε, προστασία δεδομένων πρέπει να προστατεύσουμε προστατεύσουμε τους πολίτες και όχι τους προβληματικούς ε, επιβάτες. Δηλαδή εδώ αντιλαμβάνεστε ότι αναφέρομαι στην εγκληματικότητα και στην προστασία της τρομοκρατίας. Δηλαδή δεν θα πρέπει να, ε, ε, ε, να κινηθούμε προς, προς διατυπώσεις οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν λαθασμένα. Επίσης το σημείο κινήσεως ήταν η τρομοκρατία και η σοβαρή εγκληματικότητα οπότε δεν θέλω να δημιουργήσω προβλήματα αλλά θα πρέπει όλες οι χώρες να συμφωνήσουν σε, μια έναν κοινό αποδεκτό ορισμό. Το θέμα είναι όντως διεθνός και το θέμα αυτό πρέπει να συζητηθεί ε, και διεθνώς αλλά θα πρέπει η Ευρώπη να εφαρμόσει ενιαίους κανόνες γιατί δεν υπάρχει ε, λόγος να περιπλέκουμε τα πράγματα στην Ευρώπη όταν ήδη έχουμε κάνει κάποια προεργασία. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει συντονισμός με επιτροπές, να προστατεύσουμε ε, τους πολίτες χωρίς όμως να μπορούν να επωφεληθούν της προστασίας αυτής οι σοβαροί εγκληματίες, ε, ε, διεθνής αντιμετώπιση. Αυτές είναι οι προτάσεις μου για να αποφύγω περιπλοκές όσον αφορά ε, τις χρηματικές επιπτώσεις για τις αεροπορικές εταιρείες είναι ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει και ε, θα πρέπει ε, να ρυθμιστεί με τρόπο ανεκτό και αποδεκτό. Ευχαριστώ. Η κυρία Τικάου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Καταρχάς, πρέπει να επισημάνουμε το γεγονός ότι στην Ευρώπη υπάρχουν διαφορετικές καταστάσεις στα διάφορα κράτη-μέλη όσον αφορά τα PNR. Υπάρχουν ε, κράτη-μέλη που έχουν εθνικές διατάξεις, υπάρχουν κράτη-μέλη που αυτή τη στιγμή εξετάζουν το ενδεχόμενο να εκπονήσουν συγκεκριμένε διατάξεις και υπάρχουν και χώρες οι οποίες δεν έχουν καμία διάταξη που να αναφέρεται ε, στα PNR. Γι' αυτό και οι κανόνες που εφαρμόζονται στα διάφορα κράτη-μέλη μπορούν να απέχουν μεταξύ των τη σήμερα ημέρα. Βεβαίως, όπου θα αναπτυχθούν εθνικά PNR, θα πρέπει να τηρούνται κάποιοι ευρωπαϊκοί κοινοί κανόνες. Θα συμφωνήσω με τους προλαλήσαντες ότι πρέπει να διευκρινίσουμε τους ορισμούς. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να περιορίσουμε το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας ε, σε σχέση με το πεδίο εφαρμογής που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι είναι υπερβολικά αυτά που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιδίως... Ε, όσον αφορά το χρόνο αποθήκευσης των δεδομένων. Πέντε χρόνια είναι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα ήθελα επίσης να επιστήσω την προσοχή σας ε, στο εξής. Υπάρχει μια οδηγία που αναφέρεται στην ε, διατήρηση ε, στοιχείων από τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, διατήρηση στοιχείων από, τους, από τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών εννοώ. και έγινε μεταφορά με δυσκολία στην εθνική νομοθεσία της συγκεκριμένη διάταξη. Το Ρουμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο, ε, καθώς επίσης και το Τσεχικό και το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο, θεωρούν ότι κάποιες από τις διατάξεις της συγκεκριμένη οδηγίας παραβιάζουν θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών, όσον αφορά την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, αλλά και άλλα θεμελιώδη δικαιώματά τους. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο στις συγκεκριμένες χώρες που σας ανέφερα, η εφαρμογή της οδηγίας αυτής έχει καθυστερήσει θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα ε, διότι έχει πλέον δημιουργηθεί προηγούμενο και κάθε φορά που θα συζητάμε ε, θέματα αυτά όπως τώρα που συζητάμε την οδηγία για τα PNR και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα στοιχεία των επιβατών θα πρέπει να δούμε κατά πόσον είναι απαραίτητα και κατά πόσον ε, μπορεί να γίνεται διατήρηση, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων όσον αφορά τη διαβίβαση των δεδομένων ή τα αποτελέσματα των αναλύσεων ε, ε, βάσει των δεδομένων αυτών ε, σε τρίτες χώρες θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί διότι εγώ θεωρώ ότι δεν θα μπορέσουμε να διαβιβάσουμε δεδομένα αυτής της μορφής σε τρίτες χώρες Ιδίω όταν πρόκειται για χώρε με τι οποίε η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει διμερεί συμφωνίε που να καλύπτουν επακριβώ τη συγκεκριμένη διαβίβαση. Σα το λέω αυτό διότι αναφερόμαστε σε προσωπικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν την ιδιωτική ζωή των επιβατών σε κάποιε περιπτώσει και γι' αυτό ακριβώ θα πρέπει να προστατεύονται δεόντω βάσει τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ε, γνωρίζω ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες δεν έχουν σχετική νομοθεσία ή η νομοθεσία είναι ε, πολύ πιο κάτω των ευρωπαϊκών προτύπων. Γι' αυτό ακριβώς και η διαβίβαση σε τέτοιες χώρες θα πρέπει να γίνεται μόνο σε περίπτωση ύπαρξης δημερού συμφωνίας η οποία περιλαμβάνει σαφέστατες διατάξεις και διευκρινίζει σαφώς ότι υπάρχει ανάλογη προστασία στις χώρες αυτές με την ευρωπαϊκή προστασία. Όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων, η επεξεργασία θα πρέπει να γίνεται σε ευρωπαϊκή επικράτεια. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα για το συγκεκριμένο ζήτημα και τέλος θα ήθελα να αναφερθώ στο εξή. Συμφωνώ με τους συναδέλφους που επεσήμαναν πόσο σημαντικό είναι να λάβουμε υπόψη και το κόστος κατά την εφαρμογή των συγκεκριμένων μέτρων. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα αναλάβει το κόστος. Καταρχάς, πώς θα υπολογίσουμε το κόστος, ποιο τμήμα της δαπάνης θα είναι των αερομεταφορέων, ποιο τμήμα θα είναι των κρατών μελών, ε, πώς θα υπολογίζεται, υπάρχουν τα οικονομικά μέσα για να γίνει κάτι τέτοιο. Και τέλος, κάτι εξίσου σημαντικό, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στην εξής πτυχή. Αν θέλουμε να είμαστε βέβαιοι ότι τα κράτη-μέλη δεν εφαρμόζουν εθνικά μέτρα τα οποία πηγαίνουν πέραν των ε, όσων προβλέπει η οδηγία, θα πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο ενός κανονισμού. Θα ήταν καλύτερο να υπάρχει ένας κανονισμός και θα ήθελα να απευθύνω τη σχετική πρόταση και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και στους συναδέλφους. Μήπως θα ήταν καλύτερη η επιλογή ενός κανονισμού και όχι μιας οδηγίας. Προσβλέπω στην ε, συνάντηση των σκιωδών εισηγητών και να ακούσω και τις απόψεις των συναδέλφων εκεί διότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και θα πρέπει να ε, δρούμε υπεύθυνα όταν ασχολούμαστε με τα συγκεκριμένα συγκεκριμένα θέματα. Ευχαριστώ την κυρία Τσικάου, ο κύριος Στέρξ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εξ ονόματο του Όλη Σμιτ θα μιλήσω, γι' αυτό θα σα διαβάσω ένα κείμενο στα αγγλικά. Καταρχά θα ευχαριστήσω την κυρία Λίχτεμπεργκερ, διότι έχει ε, μια ευαίσθητη προσέγγιση στα θέματα τη αναλογικότητα, της ασφάλειας και τη προστασία των επιβατών. Θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη ισορροπία, προκειμένου να μην υπάρχει υπερβολικό άχθο για του επιβάτε και τι αεροπορικέ εταιρείε και να μην υπάρχει πρόσκομα για την ελεύθερη μετακίνηση των ε, ε, επιβατών στην Ευρώπη. Μα ενδιαφέρει ο χρόνος κράτησης των δεδομένων και το γεγονός ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν ε, και για συγκεκριμένο τρόπο. Τα πέντε χρόνια είναι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ξέρω ότι το Συμβούλιο θα προσπαθήσει να επιμηκύνει ακόμα περισσότερο το συγκεκριμένο ζήτημα, γι' αυτό καλό θα ήταν να βρούμε μια κοινή θέση εδώ. 30 μέρες όμως είναι ίσως πολύ μικρό χρονικό διάστημα γιατί τότε δεν θα έχουν καμία χρησιμότητα τα PNR. Θα πρέπει επίσης να δούμε και τις συζητήσεις με τον ενδιαφερομένους για να δούμε ποιο είναι το κατάλληλο χρονικό διάστημα και να έχουμε και τη δυνατότητα επιμήκυσης της περίοδου διατήρησης ελαχίστων ε, δεδομένων ε, που θα κρατούνται ανώνυμα και τι σημαίνει ανώνυμη χρήση των ε, δεδομένων. Ορισμένες φορές το πλαίσιο είναι πολύ ευρύ, πολύ ε, ακατάλληλο στη χρήση για τα PNR και καλό θα ήταν να μην μείνει όπως έχει στην παρούσα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, όμως, τη χρήση των στοιχείων PNR για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας μπορεί να είναι πολύ στενό πεδίο εφαρμογής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για το οργανωμένο έγκλημα και την εμπορία ανθρώπων. Θα πρέπει επίσης να δούμε πώς θα καθορίσουμε τις συγκεκριμένε κατηγορίες σαφώς ε, για να μην υπάρχει καμία παρανόηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ράντμπορν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολλά από αυτά που ελέγχθησαν να με βρίσκουν σύμφωνο αλλά υπάρχουν ορισμένα άλλα θέματα που εθίγησαν και θα ήθελα να τα εξετάσω από μια διαφορετική σκοπιά από ότι η ε, νομική επιτροπή του Κοινοβουλίου στην προηγούμενη ε, θητεία και όλα αυτά αναφέρονται βέβαια στα PNR της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Υπάρχει ένα θέμα κλειδί και το θέμα κλειδί το οποίο αναφέρθη εν παρόδο είναι ο περιορισμός διότι αν όντω θέλουμε ε, να έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα γίνεται σεβαστό θα πρέπει να έχει ε, συγκεκριμένο περιορισμένο στόχο. Πρέπει να είναι περιορισμένο από πλευράς του ορισμού για τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς ε, ε, τα, για τα εγκλήματα για τα οποία μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει τα PNR και θυμάμαι στο προηγούμε, στην προηγούμενη θητεία του Κοινοβουλίου είχαμε εξετάσει μία παρεμφερή κατάσταση που ήταν το Ευρωπαϊκό Ένταλμα λήψεως και μας είχαν διαβεβαιώσει ότι θα χρησιμοποιείται μόνο σε πολύ σοβαρά εγκλήματα και βλέπουμε ότι τελικά χρησιμοποιείται ε, και ε, για την λαθρεμπορία χειριδίων που δεν νομίζω ότι ήταν το σοβαρό έγκλημα το οποίο είχαμε κατά νου όταν νομοθετήσαμε. Χρειάζεται λοιπόν ένας ορισμός των σοβαρών σοβαρών εγκλημάτων και πρέπει να ξέρουμε τι είναι τα σοβαρά εγκλήματα. Ο κύριος Στέρξ αναφέρθηκε στο εμπόριο ανθρώπων, στο εμπόριο ναρκωτικών και έχει δίκιο. Αυτά είναι σοβαρά εγκλήματα. Αλλά καθυστερεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, ε, ποιοι οργανισμοί θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία αυτά. Και αυτό που το θα ήθελα να περιληφθεί στην έκθεση αυτή είναι ε, μία δήλωση σχετικά με τις, ε, τους οργανισμούς που θα ε, εξουσιοδοτούνται να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία αυτά. Στο Ηνωμένο Βασίλειο η υπάρχει μόνο σε πολύ αυστηρή νομοθεσία ένας οργανισμός που μπορεί να το χρησιμοποιήσει, το UK Border Agency. Το αντίστοιχο θα έπρεπε να υπάρχει και αλλού. Το εάν θα μπορέσει αυτό να ισχύσει σε ολόκληρο το Σέγγεν είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζω και θα ήθελα περισσότερες διευκρινήσεις. Μετά, η περίοδος κατακράτησης των στοιχείων Βεβαίω Βεβαίως θα θέλαμε να υπάρξει μια συμβιβαστική λύση σύμφωνα με την οποία τα στοιχεία θα είναι χρήσιμα διότι διαφορετικά δεν είναι χρήσιμα σε κανέναν αλλά συγχρόνως πρέπει να εξασφανίσουμε ότι θα υπάρχει περιορισμός όσον αφορά την περίοδο όταν χρησιμοποιούνται αυτά τα στοιχεία όντως και όχι είναι παραπεταμένα σε κάποιο αρχείο. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε ένα διαχωρισμό μεταξύ του ενεργού υλικού και του αδρανούς υλικού. Ένα άλλο θέμα είναι ε, ε, ε, ένα στο οποίο διαφορώ με την κυρία Λίχτεμπέργκερ που θέλει να διαγράψει ορισμένα θέματα διότι παραδείγματο χάρη θέλει να διαγράψει το σημείο 6 που αναφέρεται με τις πληροφορίες για τις πληρωμές, την διεύθυνση διεύθυνση χρέωσης. Εάν όμως αναφερθείτε στις συνοριακές αρχές, αν κάποιος αγοράσει ένα εισιτήριο με μία πιστοτική κάρτα, ξέρει κανείς πώς έχει χρησιμοποιηθεί το, χρησιμοποιηθεί, έχουν χρησιμοποιηθεί τα χρήματα. Ενώ αν πληρώσετε τις μετρητής δεν υπάρχει αυτό το στοιχείο και πρέπει να μπορούν ε, να παρακολουθήσουν αυτές τις πληροφορίες οι υπεύθυνοι. Το ίδιο είναι ε, και τα προγράμματα των τακτικών επιβατών και των προορισμών τους οποίους ε, επισκέπτεται κανείς τακτικά. Καλό είναι να έχουμε πληροφορίες σχετικά με την μορφή ταξιδιού κατά τρόπον ώστε να μπορεί κανείς να γνωρίζει ποια είναι τα στοιχεία που μπορούν να μας, να μας δείξουν που υπάρχουν δυνητικοί, ε, δυνητικές απειλές. Επίσης, θα πρέπει ο αποδέκτης να είναι ο, υπε, οργανισμός που χειρίζεται αυτές τις πληροφορίες. Όταν λοιπόν θα κοιτάξουμε το θέμα αυτό πρέπει να δούμε ε, ποιος θα είναι ο μηχανισμός που θα ισχύσει στο τέλος στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και ο οποίος θα πρέπει να συνάδει όχι μόνο στα κράτη-μέλη αλλά και ε, με τις συμφωνίες που διαπραγματευόμαστε με τρίτες χώρες σχετικά με τα PNR γιατί θα είναι ανόητο να έχουμε ε, άλλους κανόνες για την Ευρώπη και άλλους για την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες χώρες όπως η Καναδάς, η Αυστραλία και τα λοιπά. Θα πρέπει όλα αυτά να μπουν σε ένα καλάθι. Εδώ σταματάω κύριε Πρόεδρε και ελπίζω ότι θα μπορέσω να διατυπώσω ορισμένες προτάσεις οι οποίες θα γίνουν αποδεκτές και από τον εισηγητή και από ορισμένους άλλους. Η κυρία Ντεβεράκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ την κυρία Λίχτεμπέργκερ για την έκθεση αυτή η οποία βασίζεται στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των επιβατών. Και είμαι βέβαιη και ότι η Επιτροπή Λύπε θα επικεντρωθεί στη προστασία των δεδομένων και στα σχόλια του Ευρωπαϊκού Ελεγκτή και του Οργανισμού των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να εναρμονιστούν τα στοιχεία των ε, επιβατών στις 27 χώρες μέλη και όπως είπε ο Ματιό Γκρό, αυτό θα επιτρέψει να καταπολεμήσουμε καλύτερα το διεθνές οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία. Ως μέλος της Επιτροπής Τραν θα ήθελα να επιμείνω κυρίως στο ότι η πρόταση οδηγίας δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να περιπλέξει ακόμη περισσότερο τη ζωή των επιβατών και των αεροπορικών εταιριών. Θα ήθελα επίσης όπως και προλαλήσαντε συνάδελφοι, να χαιρετήσω την πρόταση της εισηγήτριας που ζητά έκθεση για τις χρηματοοικονομικές επιπτώσεις της οδηγίας αυτής για τους επιβάτες και για τις αεροπορικές εταιρείες. Επίσης σημαντικό είναι το σύστημα συλλογής για τη μεταφορά δεδομένων να σέβεται πλήρως ε, τη διαδικασία που ισχύει σε αεροπορικέ εταιρείε. Δεν θα πρέπει να επιβάλλει οδηγία επιπλέον διοικητικό άκθο. Θα καταθέσω και σχετικέ τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Φώστερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστήσω πολύ για τις παρατηρήσεις των συναδέλφων και τις παρατηρήσεις του κυρίου Μπράντμπουρν, ο οποίος χρειάστηκε να φύγει δυστυχώς. Κάποιε παρατηρήσεις και από πλευρά μου στις ε, τροπολογίε τη κυρίας Λίχτεμπέργκερ, διότι έκανε μεγάλη προσπάθεια επί του τους. Θα πρέπει λίγο να σκεφτούμε γιατί χρειαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες και αν τις χρειαζόμαστε. Και βεβαίως ε, πότε χρειάστηκαν αυτές οι πληροφορίες για πολύ καιρό. Τα θέματα αυτά προέκυψαν ε, για το PNR επειδή είχαμε την 11η Σεπτεμβρίου ε, και υπήρχαν και βιαιότητες και περιπτώσεις στις οποίες ε, ήταν σε κίνδυνο η σεπτεμβριου και υπηρχαν και βιαιοτητες και περιπτωσεις οι οποιες ηταν σε κινδυνο η ζωη των ανθρώπων. Γι' αυτό ακριβώς χρειαστήκαμε να εξετάσουμε το ενδεχόμενο, να έχουμε περισσότερες πληροφορίες από όσες λαμβάναμε μέχρι τούδε για τους επιβάτες. Το θέμα όμως είναι ποιος πρέπει να έχει αυτές τις πληροφορίες, ποιος πρέπει να έχει πρόσβαση όταν εξετάζεται τα στοιχεία του ε, αυτά και ποιος ασχολείται με τα ζητήματα. Η... Στο Ηνωμένο Βασίλειο η υπηρεσία συνόρων έχει 27.000 προσωπικό, αλλά ελάχιστοι εξ αυτών έχουν πρόσβαση στα στοιχεία PNR και έτσι θα πρέπει να γίνεται, διότι όπως είπαμε αυτές οι πληροφορίες δεν είναι για να τις βλέπει όλος ο κόσμος και να έχει πρόσβαση σε αυτές ε, το σύμπαν. Θα πρέπει λοιπόν ε, να δούμε τι γίνεται με αυτές τις πληροφορίες. Να δούμε τώρα και κάποιες τροπολογίες. Οι 1, 2, 7 και 8 αφορούν τα σοβαρά εγκλήματα και τον περιορισμό τους. Περιορίζουμε τα στοιχεία PNR μόνο στην τρομοκρατία. Αλλά η τρομοκρατία, ναι μεν είναι βασική σημασία, αλλά υπάρχουν και σοβαρά δικήματα που ανέφερε και ο κύριος Στέρξ. Προφανώς θα χρειαστούμε καλύτερους ορισμούς, αλλά τι είναι προφανές. Ε, οι συνάδελφοι είπαν ότι πρέπει να εξετάσουμε και το εμπόριο ναρκωτικών, το εμπόριο ανθρώπων, αν υπάρχουν βιαστέ και δολοφόνοι σε αυτά τα ε, στοιχεία. Είναι προφανή ποια είναι τα εγκλήματα που μας ενδιαφέρουν εκτός και αν είμαστε τόσο ανόητοι που δεν ξέρουμε ποιο είναι το σοβαρό αδίκημα και το σοβαρό έγκλημα. Ο συνάδελφος Μπράντμπον ε, έθιξε και το εξή ζήτημα. Αν κάποιος έχει λάβει μία κλίση για παράνομη στάθμευση, προφανώς δεν είναι επικίνδυνο εγκληματίας. Πρέπει να είμαστε λίγο σοβαροί με αυτά τα ζητήματα. Δεν μπορούμε να διαγράψουμε την αναφορά στα σοβαρά ε, αδικήματα λοιπόν. Επίσης, εγώ ως κλίδα έχω να σας πω ότι δεν έχουμε καμία πρόθεση να παροπλήσουμε το σύστημα συνόρων που έχουμε αυτή τη στιγμή. Ε, είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση με τους ανθρώπους που ήρθαν στο Ηνωμένο Βασίλειο και συναντήθηκαν και με την υπηρεσία συνόρων και με άλλους ανθρώπους και μας εξήγησαν πώς λειτουργούν τα συστήματα. Είμαι βέβαιη λοιπόν ότι δεν γίνεται κατάχρηση των πληροφοριών και χρησιμοποιούνται με τον ορθό τρόπο. Μια τελευταία παρατήρηση. Υπάρχουν κάποιες τροπολογίες που αναφέρονται στο χρόνο διατήρησης ε, ε, οι 6, οι 13, οι 14 και οι 15. Όπως είπε και ο συνάδελφος Μπράτπουν, το διάστημα των 30 ημερών δεν είναι το κατάλληλο. Εάν ε, μιλήσετε με τις υπηρεσίες που ασχολούνται με την εφαρμογή της νομοθεσίας του νόμου αστυνομικές δυνάμεις και το τι κάνουν για να συλλάβουν ε, ε, εγκληματίες. Πολλές φορές ασχολούνται τρία-τέσσερα χρόνια για να βρουν τους ανθρώπους αυτούς ε, και τελικά φτάνουν στο δικαστήριο και δεν έχουν τις πληροφορίες γιατί έχει εκπνεύσει προθεσμία διατήρησής τους. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε αν μας φτάνουν τα πέντε χρόνια, μπορεί να είναι 4,5, μπορεί να είναι 5,5 τα χρόνια. Αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε είναι να πούμε ότι δεν μπορούμε να έχουμε αυτό το χρονοδιάγραμμα, διότι όπως ε, σας είπα εξαρτάται και από το αδίκημα και από το τι συμβαίνει και πόσα χρόνια διεξάγεται μια έρευνα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται ε, σε ε, χειμερή ανάρκη. Είναι τρομοκράτες που τους έχουμε σε χειμερή ανάρκη και μετά από 15 χρόνια τους ενεργοποιούμε και τους χρησιμοποιούμε. Επομένως θα πρέπει να δούμε τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Θεωρώ ότι είναι σωστό να προσπαθήσουμε να έχουμε ένα ευρωπαϊκό σύστημα να υπάρχει δυνατότητα, να υπάρχει ένα αποτελεσματικό ε, μέσο κατά των ε, ε, απειλών ασφαλείας σε υψηλό επίπεδο, αλλά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν πρέπει να τα βάζουμε όλα στο ίδιο καζάνι. Υπάρχουν και θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά θα πρέπει να είμαστε και λίγο ρεαλιστές, διότι είναι φρικτός ο κόσμος στον οποίο ζούμε κάποιες φορές και θα πρέπει να είμαστε ένα βήμα μπροστά από αυτούς που προσπαθούν να βλάψουν την όλη κοινωνία. Ευχαριστώ και πάλι την κυρία Λίχτεμπέργκερ. Κύριος Ζασάντα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αυτός που παίρνει τελευταίο το λόγο έχει πάντοτε το πρόβλημα ότι οι προλαλήσαντες έχουν πει σχεδόν τα πάντα. Βέβαια, το να αγγιθούμε την ασφάλεια είναι ένα από τα πρωταρχικά καθήκοντα για κάθε κράτος και υπάρχουν διάφορες μέθοδοι. Έχουμε την ανάλυση των ε, λειτουργικών πληροφοριών ή επιχειρησιακών πληροφοριών των μυστικών υπηρεσιών, έλλειψη στα αεροδρόμια κτλ. Σήμερα συζητούμε για την χρήση των δεδομένων των στοιχείων των επιβατών με στόχο την αποτροπή, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας αλλά και των σοβαρών εγκλημάτων. Οι συνάδελφοί μου μίλησαν για το κόστος. Σας μιλήσουμε για το κόστος. 600 εκατομμύρια ευρώ. Και σε αυτά προσθέτουμε 16 εκατομμύρια για τους ε, operators, για τους χειριστές. Τι θα πάρουμε εμείς ως αντάλλαγμα, ρωτώ την Κομισιόν. Συμφωνώ εγώ με την ε, βασική θέση της εισηγήτριας θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην τρομοκρατία. Πράγματι. Και συμμερίζομαι τους φόβους ό,τι αφορά τη χρήση των στοιχείων των επιβατών για την καταπολέμηση των σοβαρών εγκλημάτων, αλλά είναι και πολύ αόριστο όρος σοβαρό έγκλημα. Δεν ορίζεται παρκώς. Η εμπειρία μα ε, μας διδάσκει ότι μια πάρα πολύ αναλυτική ε, ρύθμιση δεν επιτρέπει πάντοτε την εκπλήρωση των στόχων για τους οποίους είχε σχεδιαστεί. Αυτό πιστεύω ότι συμβαίνει όπως με το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Αυτά έχω να πω. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω, όπως και προλαλήσατε στην κυρία Λιχτενμπέργκερ, γιατί η έκθεση η οποία έχει εκπονήσει πραγματικά ήταν πάρα πολύ απαραίτητη. Έχω τρία προβλήματα και τρεις τροπολογίες. Ε, το πρώτο σε ό,τι αφορά την αιτιολογική σκέψη 12. Η κατάσταση και εκεί και η συζήτηση μεταξύ άλλων το πρόβλημα είναι το πεδίο εφαρμογή τη οδηγία, πόσο ευρύ δηλαδή είναι το πεδίο εφαρμογή, σε τι είδου εγκλήματα καλύπτει. Και κάποιοι ομιλητέ είπαν ότι θα ήθελαν να περιοριστεί η εξολοκλήρωση τρομοκρατία. Όπω όμω είπε η κυρία Φώστερ, ε, το έγκλημα είναι έγκλημα. Είτε είναι λαθρεμπό ναρκωτικών, είτε είναι σωματεμπορία, είτε είναι ξέπλυμα χρήματο και ούτω καθεξής. Εάν λοιπόν έχουμε μια βάση δεδομένων που θα αντιμετωπίζει όλα αυτά τα προβλήματα που είναι διακρατικά, δεν σέβονται σύνορα ε, σε καμία περίπτωση αυτά τα κλίματα, αυτή την βάση δεδομένων θα πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι ωστόσο τα κράτη-μέλη μπορούν να αποκλείσουν ε, ελάσσονα αδικήματα ε, των να λαμβάνονται υπόψη από ένα κοινό ποινικό σύστημα. Μα δεν υπάρχει κοινό ποινικό σύστημα και άρα νομίζω ότι καλύπτεται η οποιαδήποτε ανησυχία μπορεί να υπάρχει και για το πώς θα διώκονται τα εγκλήματα ή τα δικήματα στα κράτη-μέλη και για το τι αδικήματα καλύπτονται. Αυτά που είπαν οι κύριοι Μπράτπορν, η κυρία Φώστερ, ε, η κυρία Ντεβεϊρά και ο κύριο Στέρξε, με βρίσκουν σύμφωνο. Και αναφέρομαι σε αυτό το, την προθεσμία των 30 ημερών. Το οποίο είναι γελίο. Να συλλέγουμε όλα αυτά τα δεδομένα, όλε αυτέ τι πληροφορίε. Και μέσα στι 30 μέρε να τα καταργούμε. Πέντε χρόνια νομίζω ότι είναι λογικό ω διαχρονικό διάστημα. Όπω είπε η κυρία Φώστερ, δεν είναι Ξαφανίζεται η τρομοκρατία. Έτσι απλά. Και στο Στρασβούργο τηρήσαμε τους λεπτούς υγιή όταν είχαν σκοτωθεί στο Λονδίνο πριν από μερικά χρόνια πάνω από 30 άτομα. Οι τρομοκράτες περιμένουν στη γωνία. Εάν δεν καταφέρουμε λοιπόν, η κυρία Φώστα μου είπε και 15 χρόνια, αν δεν κρατάμε τα στοιχεία, τουλάχιστον 5 χρόνια, δεν, δεν καταλαβαίνω. Και το τελευταίο μου σχόλιο. Τελικά, ο στόχος της πρότασης αυτής της κυρίας Λίχτενμπέργκερ είναι καλός. Το θέμα είναι όμως να βρούμε τη σωστή ισορροπία. Να έχουμε κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες. Να φροντίσουμε ότι τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για αυτό που πρέπει. πολέμηση δηλαδή εγκλημάτων ή τρομοκρατίας. Και σίγουρα να μην πέσουν σε λάθος χέρια τα στοιχεία. Καλή έκθεση γενικά, αλλά οι τρεις τομείς που προανέφερε είναι τομείς με τους οποίους διαφωνώ εντελώς πεδίο εφαρμογή, ε, η προθεσμία και ο τρόπος προστασίας των δεδομένων. Αυτά είναι απολύτως απαραίτητα για να πετύχουν οι στόχοι και πρέπει βέβαια να σεβαστούμε και το προσωπικό χαρακτήρα των δεδομένων. Πριν δώσω το λόγο στην Κομισιόν, λέει ο Πρόεδρος, και επειδή ε, τρία ήταν τα θέματα που ουσιαστικά όλοι σχολίασαν, καταλήγοντα, βέβαια ενίοτε διαφορετικά συμπεράσματα, επειδή τρόπο επεξεργασία των δεδομένων, αποθήκευσής τους δηλαδή. Νομίζω ότι εκεί θα ίσως θα πρέπει να ψηφίσουμε. Κύριε Βασιλιάδο από την Κομισιόν έχει το λόγο. Thank you very much. Uh, thank you for... Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστούμε για την πρόσκληση και μα χαροποιεί το γεγονό ότι η Επιτροπή Μεταφορών ασχολείται με το ζήτημα αυτό και έχουμε και την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυτό το σχεδιο οδηγία. οδηγίας. Υπάρχουν ένα-δυο στοιχεία τα οποία θα ήθελα να αναφέρω. Δύο τροπολογίες επικεντρώνονται αποκλειστικώς και μόνο στις εναέριες μεταφορές, ε, τροπολογίες 10 και 17. Χαιρετίζουμε και τις δύο αυτές τροπολογίες και χαιρετίζουμε και τη συνεισφορά σας ε, εδώ. Όλοι οι ομιλητές ε, και η έκθεση αναφέρονται σε ουσιαστικά σημεία της πρότασης. Και αυτά άλλωστε θα τα συζητήσει και η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, η συναδελφοί σας. Η πρόταση είναι πολύ σημαντική για την εσωτερική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι και πολύ ευαίσθητη πρόταση. Πολλές πληροφορίες ε, που αφορούν την πρόταση είναι εμπιστευτικές, ε, διότι αφορούν την εφαρμογή της νομοθεσίας και θα ήθελα να ενημερώσω την Επιτροπή σας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έχει ξεκινήσει μια διαδικασία με, τη μέλη, τα μέλη της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών που έχει κάνει δύο συνεδριάσεις ε, και συζητούν τις βασικές προτάσεις και όλα τα βασικά ζητήματα που αναφέρεστε εσείς, το πεδίο εφαρμογή, τη διατήρησή τους, ε, το καθεστώς ε, περιορισμού των στοιχείων και συζητάμε με τα μέλη της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών αυτά τα πολύ σημαντικά θέματα. Το σχέδιο έκθεσης θα τροποποιήσει βεβαίως πολύ σημαντικά το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Και βέβαια δεν θα σας εκπλήξει το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτιμούσε να ε, τηρήσει τα όσα είχε προτείνει η ίδια αρχικώς. Θεωρούμε ότι στην Ευρώπη τουλάχιστον η πρόταση χρησιμοποιείται ως επιτοπλίστων για την καταπολέμηση των σοβαρών εγκλημάτων. Υπάρχουν πολύ σημαντικά ωφέλη από τη χρήση των δεδομένων PNR για την καταπολέμηση των σοβαρών αδικημάτων και το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης ε, χρησιμοποιείται ε, ε, εκτενώς και έχει ένα περιθώριο τριών ετών και μάλιστα όλα όσα έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τούδε στον τομέα ε, της εφαρμογής του νόμου ε, είναι ε, βάση του καταλόγου που έχουμε στο Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύντριψης για τα σοβαρά δικήματα και εγκλήματα. Επομένως, ε, η καταπολέμηση του εγκλήματος βασίζεται σε αυτό. Δεν υπάρχει βέβαια κάποιος μαθηματικός τύπος για να υπολογίσουμε ποιο είναι ο κατάλληλος χρόνος για να διατηρούμε τα στοιχεία. Οι 30 ημέρες βέβαια σαφώς δεν επαρκούν. Ο μέσος άνθρωπος ποτέ δεν θα έχει ταξιδέψει σε 30 ημέρες, επομένως δεν θα υπάρχει καταγραφή ταξιδιού ε, και δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τίποτα με στοιχεία που διατηρούμε για 30 ημέρες. Τα στοιχεία που λαμβάνουμε από τις αστυνομικές ε, και δικά ε, αρχές είναι ότι τα 5 χρόνια είναι το ελάχιστο διάστημα που δέχονται. Θα προτιμούσαν πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αλλά το πενταετές διάστημα είναι το ελάχιστο χρονικό διάστημα. Και αυτό είναι και ο χρόνος που χρησιμοποιείται και σε άλλες ε, περιπτώσεις και για άλλε βάσεις δεδομένων και άλλα ε, δεδομένα τα οποία τηρούνται για στόχους ε, αστυνομική και δικαστική συνεργασίας. Γι' αυτό θέσαμε και αυτό το όριο των 5 ετών. Θα ήθελα να αφαιρθώ σε δύο θέματα τα οποία αναφέρονται εκτενώς στο σχέδιο έκθεση, αλλά δεν συζητήθηκαν σήμερα. Πρώτον, το θέμα του καθεστώτος προστασίας δεδομένων. Εμείς προτείνουμε το καθεστώς να είναι η απόφαση πλαίσιος για την προστασία δεδομένων που ασχολείται με την ε, προστασία δεδομένων στην εφαρμογή ε, του νόμου. Δια νόμου αυτή είναι η απόφαση που ισχύει. Παρά το γεγονός ότι η οδηγία 9546 μπορεί να έχει υψηλότερε προδιαγραφές ασφαλείας, εκ νόμου δεν εφαρμόζεται. Γι' αυτό ακριβώς επιλέξαμε και το καθεστώς που έχουμε επιλέξει. Τέλος, ένα θέμα που αναφέρεται επίσης και δεν αναφέρθηκε σήμερα είναι οι τροπολογίες 1 και 9 και τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη χρήση, τους χρήστες των στοιχείων PNR και η χρήση για αξιολόγηση κινδύνου σε πραγματικό χρόνο των δεδομένων. Αυτό είναι ο πυρήνας των όσων γίνονται με τα στοιχεία PNR. Εάν αφαιρεθεί το συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογή και δεν υπάρχει δυνατότητα χρήσης του PNR για αυτό το σκοπό, δεν έχουμε και λόγο χρήσης των PNR. Γι' αυτό λοιπόν καλό θα ήταν να επανεξετάσετε την άποψή σα για τις τροπολογίες αυτές. Το κόστος τώρα σαφώ είναι πολύ σημαντική πτυχή, διότι οι αερομεταφερεί ε, θα ε, έχουν σχέση με αυτή την πρόταση. έχει αξιολογηθεί τι κόστος ε, περιλαμβάνεται για τους αερομεταφερές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε και μια ανεξάρτητη μελέτη που και πάλι αξιολόγησε το κόστος. Δεν πρόκειται λοιπόν για μια τυχαία άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι εμπειρογνώμονες μας πρότειναν το συγκεκριμένο ζήτημα. Το κόστος είναι σημαντικό, είναι ουσιαστικό, αλλά θα πρέπει επίσης να επισημάνουμε ότι παρά το γεγονός ότι μπορεί να είναι υψηλό το αρχικό ποσό, είναι λιγότερα από 10 cents του ευρώ ανά επιβάτη και αυτό είναι με υπολογισμό με, την με το υψηλότερο δυνατό κόστος και τη διαβίβαση των δεδομένων. Στην πράξη λοιπόν το κόστος δεν είναι τόσο υψηλό όσο φαίνεται εκ πρώτης όψεως. Τέλος, θα ήθελα να σημειώσω ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα η έκθεση αναφέρεται στη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Συμβουλίου και δίνει και ένα σύνδεσμο για μια ιστοσελίδα την οποία μπορείτε να κατεβάσετε το συγκεκριμένο, ε, τη συγκεκριμένη γνωμοδότηση. Δύο στοιχεία εδώ. Καταρχάς αυτή η γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Συμβουλίου αναφέρεται ή μάλλον διορθώνει ομιλήτρια. Αυτή η γνωμοδότηση είναι εμπιστευτικό έγγραφο, ε, καλύπτεται από ε, νομική εμπιστευτικότητα και έχει διαρρεύσει παρανομω στον τύπο και τώρα διατίθεται online. Ε, καλό θα ήταν λοιπόν να διαγραφεί αυτή η αναφορά ε, με την παραπομπή στη νομική γνωμοδότηση. Υπάρχει νομική εμπιστευτικότητα για όλα αυτά τα θέματα και καλό θα ήταν να μην αναφέρεται τουλάχιστον αυτό εδώ. Κυρία Λίχτεμπεργκερ, θέλετε να πείτε κάτι επιπλέον εδώ. Όχι, δεν διέρευσα εγώ το έγγραφο αυτό διότι το έσκησα. Ε, μπορώ όμως να μιλήσω γερμανικά, λέει η συγγήτρια. Καταρχήν, σχετικά με τις αντιρρήσεις ε, οι οποίες διατυπώθησαν από τους διάφορους και όδης θα ήθελα να πω το εξής. Στη συζήτηση αυτή υπάρχει πάντοτε μία σύγχυση μεταξύ της παρακολούθησης μεμονωμένων περιπτώσεων που είναι εφικτή με την ε, δικαστική συνεργασία και όπου σε μεμονωμένες περιπτώσεις υπάρχει η αμοιβαία δικαστική βοήθεια και αυτό είναι σαφές. Δεύτερον, τα στοιχεία όλων των ε, επιβατών ε, θέλουν ορισμένοι να μπορούν να τα ερευνούν διότι μπορεί να σκέφτεται ότι ένας που πηγαίνει από εδώ είναι έμπορος ναρκωτικών και κάποιος που πηγαίνει στην Αιδία είναι τρομοκράτης. Δηλαδή ε, υπάρχουν, ε, θεωρούν ότι ε, οι εγκληματίες πηγαίνουν σε συγκεκριμένους προορισμούς ενώ μπορεί να πάει κανείς στη Γουατεμάλα για άλλους λόγους εκτός τα ναρκωτικά και στην Ινδία ή στο Πακιστάν για άλλους λόγους και όχι υποχρεωτικά λόγω της τρομοκρατίας. Οπότε ε, δεν είναι δυνατόν έτσι συλλήβδη να μπορεί κανείς να κοιτάζει και να αναλύει όλα τα στοιχεία και εκεί δημιουργείται και το πρόβλημα το οποίο ανέφεραν ορισμένοι σχετικά με τη διασύνδεση με τη σκοπιμότητα. Δηλαδή αν τα κράτη-μέλη μπορέσουν να καθορίσουν τι θεωρούν σαν ένα σοβαρό έγκλημα, αν έχουμε διαφορετικούς ποινικού κώδικες τότε θα έχουμε πρόβλημα διότι το κάθε κράτος θα είναι ελεύθερο, παραδείγματος χάρη, να περιλάβει ακόμη και τις ε, ε, τα παραπτώματα οδικής κυκλοφορίας ε, στο, στα εγκλήματα. Εγώ θα ήθελα όμως να υπάρχει ένας έλεγχος όπου είναι ε, μία σοβαρή περίπτωση, είναι θέμα αναλογικότητος. Εάν μπορώ να έχω ανα πάσα στιγμή μπροστά μου όλα τα στοιχεία όλων των Ευρωπαίων πολιτών ε, με τους αντιστοίχους αλγορίθμους τότε βέβαια ε, θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και το κόστος το οποίο αυτό θα συνεπάγεται. Θεωρώ ότι είναι πολύ βασικό. Εάν αποφασίσουμε να ε, χρησιμοποιήσουμε τέτοιους μηχανισμούς να τους συνδέσουμε με τους στόχους στόχους μας. Π.χ την τρομοκρατία. Ορισμένοι συνάδελφοι ε, ήδη ανέφεραν τι άλλες αξιόπινες πράξεις θέλουν να συμπεριλάβουν, αλλά με το τωρινό καθεστώς, όπως εγώ ερμηνεύω την ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το σύστημα αυτό για πάρα πολλά πρόγραμμα, διότι ε, σε εδώ και τρία χρόνια υπάρχουν μακροί κατάλογοι από τα κράτη-μέλη όπου τα εγκλήματα περιλαμβάνουν μακριές λίστες ε, που μπαίνουν τα πάντα. Δεύτερον, σχετικά με την, ε, προθεσμία ε, κατακράτησης και αποθήκευσης των στοιχείων. Ορισμένοι είπαν ότι οι 30 μέρες δεν είναι επαρκής. μίλησε η κυρία και έχω και Γερμανούς συναδέλφους οι οποίοι διαφωνούν και πρέπει να πούμε ότι σύμφωνα με τις δικαστικές αποφάσεις πρέπει να δούμε τι είναι ακόμη εφικτό διότι υπάρχουν χώρες που όπως σας είπα δεσμεύονται από αποφάσεις των συνταγματικών δικαστηρίων όπως η Γερμανία παραδείγματο χάρη. Οπότε ε, υπάρχει η υποψία της ε, κατακράτησης ε, ε, προσωπικών δεδομένων. Και, λοιπόν, αν μιλάμε για αποθήκευση πρέπει να ξέρουμε ότι εδώ πρόκειται για στοιχεία τα οποία θα είναι ανωνυμοποιημένα. Αλλά όταν απλώς έχουν καλυφθεί σημαίνει ότι η ιεραρχία τα έχει μετακινηθεί κατά μία βαθμίδα που κατ' εμέ δεν προσφέρει επαρκή προστασία σε σχέση με τις πράξεις. Όσον αφορά τα στοιχεία για τις ε, πιστοτικές κάρτες ε, πρέπει να δούμε εάν καταγράφεται κάποιος ο οποίος πληρώνει μετρητής άρα είναι ύποπτος ή αν ε, πληρώνει και με πιστοτική κάρτα και αν παρακρατώ και αποθηκεύω όλες τις πληροφορίες για όλες τις πληρωμές με ε, πιστοτικές κάρτες. Είμαι στη διάθεσή σας να ξανασυζητήσουμε το θέμα αυτό. Προσβλέπω σε μια επικοδομητική συζήτηση, αλλά πιστεύω ότι ήδη στο σημείο αυτό καλό θα ήταν να λάβουμε υπόψη μας ότι δεν πρέπει να κοιτάξουμε όλη τη διαδικασία ποινική διώξεως, αλλά να μπορεί κανείς να ε, επεξεργαστεί και να ελέγξει τα στοιχεία ενός μεμονωμένου επιβάτη, να υπάρξει μία ανταλλαγή με μία τρίτη χώρα όπου χάνουμε τον έλεγχο της χρήσεως αυτών των στοιχείων περαιτέρω. Και γι' αυτό αγαπητοί συνάδελφοι ξανασκεφτήκα το διότι ε, είναι θέματα διεθνών σχέσεων, είναι ε, λεπτά θέματα που έχουμε συζητήσει πολλές φορές και εκεί δημιουργούνται δυσκολίες. Είναι κάτι που δεν μπορούμε να ελέγξουμε, δεν μπορούμε ε, να υπαγορεύσουμε στις νομένες Πολιτείε αν έχουν στοιχεία σχετικά με τους Ευρωπαίους πολίτες τι θα τα κάνουν και τι όχι και οι κίνδυνοι να φτάσουν όλο και περισσότερο στοιχεία στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξάνονται συνέχεια γιατί οι ΗΠΑ μας ζητούν όλο και περισσότερα. Αυτά είναι οι απαντήσεις μου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και επιπλέον, εάν έχω λάβει αυτό το έγγραφο απλώς και μόνο διότι παρουσιάστηκε στο διαδίκτυο, δεν ε, θεωρώ ότι μπορούμε απλώς να το διαγράψουμε σαν να μην υπήρξε ποτέ διότι όπως σας είπα συζήτησα με συναδέλφους ε, το, της Επιτροπής Ελευθεριών διότι είχαμε συμφωνήσει ότι θα ανταλλάσσουμε τις πληροφορίες που οδηγούν στη λήψη των αποφάσεών μας και αυτό που εγώ επιζητώ είναι να έχουμε ένα σωστό ορισμό της εγκληματικότητας διότι θα δείτε στα, ε, στις εθνικές νομοθεσίες ότι υπάρχουν πάρα πολλές διαφορές και θεωρώ ότι δεν είναι δυνατό να προχωρήσουμε με όλες αυτές τις συμπτώσεις. Δεν θέλω να διατυπώσω συγκεκριμένες προτάσεις αυτή τη στιγμή, θέλω να συνεχίσουμε να συζητάμε και προσβλέπω στις προτάσεις που θα μου υποβάλλετε. Σε ευχαριστώ. 7 Σεπτεμβρίου λίγη προθεσμία κατάθεση τροπολογιών και στην Επιτροπή μας θα ψηφίσουμε τον Οκτώβριο. Σας ευχαριστώ. Και περνάμε στο επόμενο θέμα, Σύμβαση των Αθηνών, που είναι δικό μου σχέδιο έκθεση. Να πω λίγα πράγματα εισαγωγικά. Ελπίζω να το εκπαιρεώσουμε γρήγορα το θέμα. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι η προσχώρηση στη Σύμβαση των Αθηνών είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει πολύ το Κοινοβούλιο, μια μακρά διαδικασία. Από το 1975 μιλάμε, αλλά το πρωτο... για το πρωτόκολλο του 2002, ουσιαστικά αυτό το οποίο λύνει διάφορα στήματα τα οποία δεν καλυπτόντουσαν από την ίδια τη σύμβαση, όπως είναι η ευθύνη ε, των ε, μεταφορέων κτλ. Από τον Απρίλιο του 2009 τα ουσιώδη ζητήματα του πρωτοκόλλου έχουν περιληφθεί, ε, αποτελούν πλέον ε, κοινοτικό δίκαιο. Υπάρχει ειδικό κανονισμό για την ευθύνη των μεταφορέων ε, επιβατών δια σε περίπτωση ατυχήματο. Μετά την έγκριση του κανονισμού αυτού, η Κομισιόν υπέβαλε ενημερωμένη, επικαιροποιημένη πρόταση ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει συμβαλόμενο μέρο τη σύμβαση. Όπω με κάθε διεθνή συμφωνία, απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου για την ολοκλήρωση τη συμφωνία. Τώρα, κανονικά, η σύμφωνη γνώμη δίνεται στο πλαίσιο μιας σύσταση, αλλά στην περίπτωση αυτή έχουμε το εξή ασύνηθες. Μετά την απόφαση του Συμβουλίου να εγκρίνει δύο συστάσει. μία από την Επιτροπή μας που βασίζεται στο άρθρο 100 για τις μεταφορές και δεύτερη σύσταση από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Η δεύτερη αυτή γνωμοδότηση καλύπτει τα άρθρα 10 και 11 του πρωτοκόλου που έχουν να κάνουν με τη δικαστική συνεργασία σε ζητήματα αστικού δικαίου, εμπορικά ζητήματα και εφαρμογή επιβολή των αποφάσεων. Έγινε αυτό ο διαχωρισμό τη νομική βάση γιατί οι διατάξει τη συνθήκη για την ε, δικαστική συνεργασία έχουν, ε, ε, έχουμε εκεί την εξαίρεση της δανεια opt opt-out. Η Δανία βέβαια θα δεσμεύεται από τα άρθρα αυτά το 10 και το 11 ως ένα ξεχωριστό συμβαλόμενο μέρος. Τώρα η τροποποίηση του κείμενου της, του κειμένου συμφωνίας δεν είναι παραδεκτές, άρα μόνο μπορεί κανείς να απορρίψει την όλη συμφωνία, εάν δεν τον ικανοποιεί. Προτείνω το εξής. Εάν κάποιοι θέλουν να απορρίψουν μέχρι τις 14 Ιουλίου στις 3 το μεσημέρι μπορούν να το πράξουν. Είχαμε προτείνει και ελπίζαμε να ψηφιστεί αύριο στην Επιτροπή μας η αλλά δυστυχώς δεν θα καταστεί δυνατό αυτό. Η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων δεν έχει συζητήσει ακόμη το θέμα, εξού και η ψηφοφορία τη επιτροπή Μεταφορών θα γίνει τον Οκτώβριο. Θέλει κάποιος να σχολιάσει, κύριος Κόζα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να επιβεβαιώσω ότι καταρχάς δεν θα μακρηγορήσω και θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε πολύ σύντομα με το σημείο αυτό στην ημερήσια διάταξη. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Συμφωνώ μαζί σας, εξ ονόματος του ΕΛΚ και από πλευράς μου βεβαίως προσωπικά μπορώ να σας πω ότι συμφωνώ με την έκθεση. Ε, είναι ε, σημαντικό το ζήτημα αυτό για να ενισχύσουμε και τα δικαιώματα των επιβατών και όπως είπε και ο ίδιος ο συζητητής έχει πάει μακριά η βαλίτσα και πρέπει κάποια στιγμή να ολοκληρωθεί αυτό το ζήτημα. Βρισκόμαστε και σε μια κρίσιμη καμπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βρεθεί εντός αυτού του ζητήματος. Θα ήθελα εδώ να σας αναφέρω και κάποιες σκέψεις μου δεν είναι σημαντικό μόνο να εγκρίνουμε την ε, συμφωνία, αλλά θα πρέπει να ελέγξουμε και ότι θα εκτελείται στο μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ασκήσει πιέσει ώστε να εφαρμόζεται ορθώ στο μέλλον. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Κόζα, ο κύριος Κόλσον από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Λίγα λόγια μόνο. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για την έκθεση που εκπονήσατε, να ευχαριστήσω και τον ε, κύριο Κόζα που μίλησε και το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι όταν ε, επικυρωθεί από τα κράτη-μέλη και την Ένωση η σύμβαση αυτή, θα μπορεί πολύ γρήγορα να εφαρμοστεί διεθνώ πλέον η σύμβαση δεδομένου του βάρους που έχει η Ένωση, που έχουν τα κράτη-μέλη μα στην προκειμένη περίπτωση. Ένα τελευταίο σημείο. Θέλουμε το συντομότερο δυνατό να γίνει αυτό πριν τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός 392 ε, του 89. Και θέλουμε να εγκριθούν το συντομότερο δυνατόν, ε, θέλουμε να εγκριθεί το συντομότερο δυνατό και πριν το τέλειο του 2011 το κείμενο της σύμβασης. Είπατε ότι η Δανία σε ό,τι την αφορά θα επικυρώσει ξεχωριστά τη σύμβαση. Ευχαριστώ. Okay, thank you very... Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Επομένως ολοκληρώσαμε με τη σημερινή ημερήσια διάταξη. Ε, θα περάσουμε τώρα απευθεία στην εδρία των συντονιστών. Παρακαλώ όσου δεν έχουν σχέση με τις συνεδρίες των συντονιστών να αποσυρθούν από την αίθουσα ησύχως. Ευχαριστώ.